Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ συγγήτριας και οδών ε, των πολιτικών ομάδων συνέχισαν και χθες το βράδυ και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε όπως είπαμε χθες το απόγευμα, να ολοκληρώσουμε το σύνολο της ψηφοφορίας σήμερα το μεσημέρι. Καταλαβαίνω λοιπόν, ε, βεβαίως δεν υπάρχει συμφωνία επί όλων των σημείων, αλλά εν πάση περιπτώσει η ψηφοφορία δίνει ακριβώ αυτή τη δυνατότητα να ληφθεί μια απόφαση βάσει της πλειοψηφίας. Ωραία λοιπόν, όπως το είχαμε προβλέψει χθε, θα προτείνω να ξεκινήσουμε με μια ψηφοφορία που δεν είναι ψηφοφορία του προϋπολογισμού, αλλά είναι η ψηφοφορία του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση για την απόφαση, νομικά έτσι αποκαλείται απόφαση, σε σχέση με τις εγγύησεις δανείων που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να χορηγήσει εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής μας είναι ο Ιβαλοκάλφιν, αντιπρόεδρος, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σήμερα και γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει πολύ ενεργά χώρα στην εθνική πολιτική της χώρας του αλλά θα θυμάστε ότι μας μίλησε σχετικά κατά επανάληψη. Υπήρξε ο τριμερής διάλογος που ήταν ιδιαίτερος δύσκολος αλλά τελικά επικοδομητικός και είχε μια θετική έκβαση και συμμετείχε η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Και τελικά κατέληξε σε μια πολιτική συμφωνία και σήμερα πρόκειται για μια ενιαία ψηφοφορία προκειμένου να επικυρωθεί η συμφωνία η οποία ε, επετεύθη ε, εξ ονόματός μας από τον Ιβάλλο Κάλφιν. Ε, βάλω λοιπόν στην ψηφοφορία τη Επιτροπή Προπολογισμών την επικύρωση τη συμφωνία του Κοινοβουλίου, τη κατάθεση του Κοινοβουλίου σε αυτό το σχέδιο απόφαση. Υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ. Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ. Κατά. τρει αποχέ. Ευχαριστώ λοιπόν. Η σύσταση λοιπόν συνεπώς εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν. Άρα στη βάση αυτή θα συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε στις τροπολογίες για το προϋπολογισμό και όπως συμφωνήσαμε χθες θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει στη σελίδα 149 που αντιστοιχεί στην κατηγορία 3β. 3β. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας. Έχετε πει στην ηλεκτρονική σας κάρτα. Είσαστε έτοιμοι. Και αυτή λοιπόν σελίδα 149 είναι οι προπαρασκευαστικές ε, δράσεις, θα τις ψηφίσουμε λίγο αργότερα. Η πρώτη τροπολογία είναι 4196 ε, του κυρίου Χάρτον. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, για την 44-76 υπάρχουν μόνο σχόλια. Ο συγκριτής είναι υπέρ. Κατά, υπέρ, συγγνώμη, κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Οι πράσινοι απέχουν, εγκρίνονται τα σχόλια. Η επόμενη γραμμή. Υπάρχουν δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. 41-99. Ε, Η συγκέντρια είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η επόμενη ε, γραμμή ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα έχουμε και πάλι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Η πρώτη τροπολογία είναι 4192 του κυρίου Χάρτονγκ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 230 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καθώς και οι δύο επόμενες τροπολογίες που έχουν το ίδιο ποσό 41.05 του κυρίου Χάγκλουντ θα πρέπει να ψηφιστούν τα σχόλια και μου λένε ότι το ΕΛΚ έχει μια ε, προφορική τροπολογία. Είναι η συγγήτρια. Τι μας ε, προτείνεται. Τι μας... Ναι. Allora, l'emendamento orale è l'inserimento dopo la parola training e prima della parola language. Εκεί πάνω από τη λέξη language αυτές τις φράσεις πρέπει να μπει χρήση όλων των ε, γνωστών γλωσσών ως στα μέσα εκπαίδευσης. Μάλλον ως μέσο εκπαίδευσης. Uh, uh, και ένα άλλο κομμάτι που είναι προσαρτημένο στην κατάλογο ψηφοφορίας και μπορώ να σας το διαβάσω. Και είναι μια προσθήκη που προτείνεται σε αυτή την ίδια αλλαγή των ε, παρατηρήσεων. Μπορώ να σας το διαβάσω ή, ε, αν θέλετε, είναι αρκετά μακροσκελής. Λέει, τμήμα αυτών των κονδυλίων θα πρέπει να αφιερωθεί στην χρηματοδότηση ε, των θεάτρων μειονότητας. Το σλοβενικό ε, θέατρο της Τεριέστης θα πρέπει να κάνει το φεστιβάλ στην Τεριέστη και να ανταλλάξει τις ε, παραγωγές με τα άλλα μειονοτικά θέατρα. Θα πρέπει αυτό να παρέχει νέες ευκαιρίες για την ευρύτερη αναγνώριση και εκτίμηση και αναγνώριση των των μειονοτικών θεάτρων καθώς και το μόνιμο ε, θέατρο, το σλοβενικό θέατρο της της. Θα πρέπει να δώσει ε, βάση για τις ε, γλωσσικές μειονότητες, τον πολιτισμό τους και να τις αξιοποιήσει. Σας ευχαριστώ. Τα, οι παρατηρήσεις θα τροποποιηθούν με την εισαγωγή στο πρώτο τμήμα της, ε, της φράσης χρήσης των γλωσσών των μειονοτικών ως ε, εκπαιδευτικού μέσου και έπειτα την προσθήκη αυτού του κομματιού που σας διάβασα, το οποίο περιλαμβάνεται στα ε, κείμενα που έχετε πάρει ως προσάρτημα στην τροπολογία 4905. Μάλιστα, αυτές οι δύο προφορικές τροπολογίες ε. έχουν το ίδιο σχόλιο λοιπόν, αυτές οι δύο προφορικές τροπολογίες και αφορούν κάπω διαφορετικέ πτυχέ. Μπορούν να αποβληθούν από, κοινού σε ψηφοφορία, όχι. Άρα λοιπόν, πρώτη τροπολογία, προφορική τροπολογία, η ένταξη τη χρήση των ε, ε, γλωσσών που κινδυνεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά Δύο αποχές. Αυτό το πρώτο τμήμα συνεπώς εγκρίνεται. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο τμήμα, ε, τμήμα αυτών των κονδυλίων θα πρέπει να φερθεί κλπ. Υπέρ. Κατά. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. 32 παρόντες με μία κάρτα Λοιπόν, πέρα στις ψηφοφορίες, για αυτό το δεύτερο τμήμα, 15 ψήφοι υπέρ, 16 κατά, άρα αυτό το δεύτερο τμήμα δεν εγκρίνεται, απορρίπτεται. Ωραία λοιπόν, στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Κληρονομιά, το σήμα για την Ευρωπαϊκή Κληρονομιά, πιλωτικό πρόγραμμα. Τα πολυμέσα 2007, η τροπολογία του κυρίου ε, Χάρτονγκ, ε, 93, η τροπολογία υπαριθμών 93. Ε, το artist mobility, η κινητικότητα των καλλιτεχνών. Ωραία. Ο κύριος Ζαβέλ ε, κοιμάται. Ε, 41-93 του κυρίου Χάρτονγκ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Η, η 46 92, ναι. 80 ε, 46 ε, υπέρ κατά 231 η συγκεκριμένη υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά κατά οι σοσιαλιστές είστε υπέρ αποχές οι 231 ε, εγκρίνεται Ωραία λοιπόν. Θα περάσουμε τώρα στην περίφημη κατηγορία τα ειδικά ετήσια προ, ε, ε, ε εκδηλώσεις. Υπάρχει μια συμβαστική τροπολογία η οποία καλύπτει 7-8 τροπολογίες όσον αφορά τα ποσά. Που τα καλύπτει όλα. Λοιπόν, όλα τα special annual events. Ε, όσον αφορά τα ποσά, έχουμε μια συμβαστική τροπολογία. Στη βάση των ποσών, τα οποία είναι 1.600.000 ε, 700.000 σε υποχρεώσεις και ένα 700 σε πληρωμές. Ωραία, λοιπόν, ποιος είναι υπέρ του συμβασμού κατά αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές, άρα συμφωνούμε επί των ποσών. Υπάρχουν κάποια σχόλια, υπάρχουν κάποια σχόλια. Υπάρχει κάποιο σχόλιο για το 60. Ποιος είναι υπέρ για την 60. Υπέρ. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού, unblock. Συγγνώμη, όχι είναι πιο απλό. Άρα λοιπόν υποβάλλεται το σχόλιο από κοινού, unblock. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ο κύριος Χάρτον. Αποχές. Εγκρίνονται συνεπώς τα σχόλια. Συγχαρητήρια. Σύμφωνα. Εν περιπτώσει λοιπόν. Όσον αφορά τις ειδικέ αιτήσει εκδηλώσει, έχει ρυθμιστεί το θέμα. Αλλά εν τω μεταξύ ο κ. Ζαβέλ ξύπνησε και ε, δεν ήταν αυτό που κοιμόταν, εγώ ίδιο ίδιος κοιμόμουν, συγγνώμη λοιπόν. Και πάμε στη σελίδα 150 για την ε, τη σήμανση για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, το σήμα ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Ξεχάσαμε ε, να ψηφίσουμε τη 4192 του κυρίου Χάρτογκ. 41-92 υπέρ του κυρίου Χάρτονγκ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία, αλλά έπρεπε να ταθεί σε ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα λοιπόν θα επανέλθουμε στην 153 του αγγλικού κειμένου. Εδώ έχουμε πιλωτικά προγράμματα, Γερνάω τη σελίδα και... Ωραία λοιπόν, στη γραμμή Νεολαία εν δράση, Youth in Action. Σας προτείνω να ψηφίσουμε καταρχήν την τροπολογία που αντιστοιχεί στη συμβαστική τροπολογία 174 ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. 174. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν καταρχήν τα ποσά και στη συνέχεια θα δούμε τα σχόλια. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές η 174 λοιπόν, όσον αφορά τα ποσά, γκρίνονται όλες οι άλλες, καταπίπτουν. Όλες οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν, δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε. Αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε τα σχόλια για την 174. είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές, άρα τα σχόλια εγκρίνονται επίσης. Και θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή, η 238. Η είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Ευχαριστώ αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη γραμμή, η 748 των πρασίνων, η είναι κατά. Υπέρ. Η πράσινη. Κατά υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. Η 239 υπέρ. Ε, η σύγκριτρα είναι υπέρ. Κατά η συντηρητική και ο κύριος Χάρτονγκ. Αποχές ευχαριστώ εγκρίνεται. Θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 44-77. Η σύγκριτρα είναι κατά. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται οι ενέργειες των πολυμέσων. Υπάρχουν ε, τροπολογίες για τα ποσά καταρχήν. Μου λένε ότι υπάρχει ένα συνολικό συμβιβασμό ο οποίος τα καλύπτει όλα. Άρα λοιπόν που αφορά τα αποθεματικά. Το αποθεματικό. Για το σύνολο. Μιλώ για μια συμβαστική τροπολογία της εισηγήτριας. Μια δέσμεση 26 εκατομμύρια 900.000 και σε, πέιμα, ε, σε πληρωμές 24 εκατομμύρια 600.000. 4 ε, εκατομμύρια 500.000 μπαίνουν στο αποθηματικό. Αυτό όσον αφορά τα ποσά. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε αυτά τα ποσά. Ποιος είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Ωραία λοιπόν για τα ποσά και το, το αποθεματικό. Υπάρχει προπόθεση να καταργηθεί το αποθεματικό σε ένα σχόλιο υπέρ. Συμβαστική τροπολογία. Κατά, αποχές, ε, προφανώς πρόκειται για την ίδια πλειοψηφία εδώ. Ωραία λοιπόν, άρα... Ωραία λοιπόν, ε, θα περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη σελίδα. Ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σας ενημερώνω ότι αν για, αυτό το, για αυτή την κατηγορία ξεπεράσουμε το σχέδιο προπολογισμού, θα ξεπεράσουμε το περιθώριο για, όλη, για την κατηγορία αυτή. Αυτό είναι ο λόγος για την οποία για την τροπολογία υπαριθμών 221 και τις υπόλοιπες που ακολουθούν και που είναι ταυτόσιμες, η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές, άρα απορρίπτεται ομόφωνα. Αντιθέτως θα πρέπει να ψηφίσουμε τη θέση αποδειγματικό. Όχι. Καταπίπτει το σύνολο. Ωραία λοιπόν. Άρα... Okay. Alors, euh, Συνέχεια έχουμε πιλωτικά προγράμματα. Ε, κέντρα μετάδοση πληροφοριών. 4602 της κυρίας Βόρτμαν. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 4286 του Γκάιερ. Η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Ο κύριος Γκάιερ. Κατά. Όλοι οι άλλοι. Λυπούμε αγαπητέ συνάδελφοι, απορρίπτεται η τροπολογία. Υπάρχει, υπάρχουν κάποια σχόλια 351, η συγκεκριμένη είναι υπέρ. Ποιο άλλο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται τα σχόλια. Και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Okay, bon. Alors, je soumets... Ωραία λοιπόν, άρα η 350, ψηφίζουμε τη 350, δημιουργία μιας νέας γραμμής. Pardon. Oui, εισηγήτρια, τι μας προτείνετε για την 350? Θα πρέπει να ψηφίσουμε μπλοκ από κοινού ή χωριστά. Παρακαλώ. Το 350 έχει μπει εδώ από λάθος. Ε, θα πρέπει τύπης να, τα ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε και για τις δύο, αλλά είναι ταυτόσιμες. Τι θα πει μαζί να τις ψηφίσουμε, δηλαδή την 350 της γραμμής 02 350 της γραμμής 0201 που θα παραμείνουν σε αυτή τη γραμμή και μου λένε ότι υπάρχει πιο κάτω το 352. Όχι, το δεύτερο τμήμα του 350-002 που αν εγκριθεί θα, θα μπει στην κατηγορία 5 Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού αυτές τις τρεις. Καταλάβατε όλοι. Εγώ δεν κατάλαβα, αλλά εσείς σίγουρα καταλάβατε. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Λοιπόν, οι δύο πρώτες τροπολογίες θα παραμείνουν σε αυτή τη γραμμή και σε αυτή την κατηγορία 3β, ενώ η τελευταία θα εγγραφεί στην κατηγορία 5. Ωραία, τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ε, ε, 10.05 της ΓΚΟΕ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 46.16 της κυρίας Βέρτμαν. Η είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 352 για θέση αποθεματικό. Αφορά τα ποσά. Με θέση αποθεματικό. Ωραία. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στη 4199 του κυρίου Χάρτογκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γυρνάω τη σελίδα. Η Ευρώπη για τους πολίτες. Έχουμε και άλλη μια τροπολογία του Χάρτον 42.00. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 347. Η είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και συνεπώς η 747 καταπίπτει. Τώρα. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, τον οίκο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών. Εδώ μια τροπολογία του κυρίου Χάρτονγκ, 4201, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, στη συνέχεια έχουμε μια προπαρασκευαστική ενέργεια, η τροπολογία παριθμών... Α, ε, συγγνώμη, 4478, ε, ναι, του κ. Βαντάλεν έχει αποσυρθεί. Έχουμε μια άλλη προπαρασκευαστική δράση στη συνέχεια, 4203 του κυρίου Χάρτονγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ο κύριος Βάντελεν καταπίπτει. Η 468 είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η, τροπολογία της κυρίας Χάου εγκρίνεται επίση. Τώρα, 4203 του κυρίου Χάρτουμ, τις επόμενες κατηγορίες, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Η Βαντάλεν καταπίπτει εκ νέου. Τώρα θα περάσουμε στη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας. Υπάρχουν σχόλια εδώ του κυρίου Λάσλο Σούριαν που η εισηγήτρια απορρίπτει. Ποιος είναι υπέρ όμως των σχολείων. Κατά. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, η 4769 ψηφίστε. Υπάρχουν τρεις που κοιμούνται ακόμα. Το στο χειρότερο για αυτούς λοιπόν. Πέρα της ψηφοφορίας. 15 υπέρ 19 κατά. Τα σχόλια του κυρίου Σουριάν απορρίπτονται. Τώρα θα περάσουμε 4204 του κυρίου Χάρτογκ. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές απορρίπτεται. Και πάλι 4489 καταπίπτει. 4204 του κ. Χάρτονγκ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 467 της Επιτροπής Περιβάλλοντος η είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. η πράσινη την καταψήφισαν αλλά είναι σε μια ψηφία η Γιούτα, της ε, καταπίπτει. Η 43-44 της κυρίας Λεπάζ αφορά μια θέση σε αποθεματικό συγκεκριμένο είναι κατά υπέρ. Κατά. Οι υπόλοιποι αποχές, άρα απορρίπτεται τώρα στη συνέχεια ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα το ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την 741 των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν. Και τελειώσαμε τώρα με την κατηγορία 3β. Και μπορούμε να φτάσουμε στην ενδιαφέρουσα κατηγορία 4. Προς μεγάλη χαρά της Αντιπροέδρου που έχει πολύ καλή διάθεση σήμερα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε από κοινού καταρχήν τα ποσά. Έχετε όλοι τους πίνακες του συμβαστικού, οι πίνακες των συμβαστικών τροπολογιών βρίσκονται στο επιπλέον ε, ντοσιέ σε μια σελίδα που δεν είναι αριθμημένη. C'est un tableau uniquement des chiffres. Πρόκειται για ποσά. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που περιλαμβάνουν ποσά και σχόλια. Θα ψηφίσουμε τα σχόλια σειρά προς σειρά στη συνέχεια, μετά. Όσον αφορά τα ποσά, τα ψηφίζουμε όλα από κοινού. Υπάρχει μια πολιτική συμφωνία για, τις 100, για να συνδράμουν τις 183 χώρες που εκπροσωπούνται στα Ηνωμένα και την Παλαιστίνη. Λοιπόν, ε, υποβάλλω αυτά τα ποσά, τον πίνακα των ποσών, σε ψηφοφορία, ε, υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά, αποχές, η πράσινη και η γκουε. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν εγκρίνονται τα ποσά. Και θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά την εισηγήτρια και τις πολιτικές ομάδες για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Ωραία λοιπόν, άρα θα ψηφίσουμε, έχουμε ένα ξεχωριστό χαρτί, αλλά πρέπει να γίνει γραμμή προς γραμμή τα σχόλια. Αυτό θα κρατήσει λίγο. Η τροπολογία 536 και οι δύο ταυτόσιμες τροπολογίες είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ, κατά. Οι φιλελεύθεροι συντηρητικοί και ο Χαρτόγκ, αλλά μειοψηφούν. Άρα εγκρίνονται αυτές οι ταυτόσιμες τροπολογίες. Η 86 του κυρίου Χάρτογκ, η συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 56 de Monsieur Σουριαν, Le rapporteur est pour. Pour. Contre. Abstention. Adopté. Αποχές εγκρίνεται. Οι δύο μεγάλες ομάδες είναι υπέρ. Ε, η 45-26 Επιτροπή Απασχόληση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 1052 της Γκουε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 4631 επίσης της Γκουε υπέρ ο κύριος Πόρτας, κατά, η λυπή, αποχές, απορρίπτεται. Η 43-32 του κυρίου Μπουσάτιλ, υπέρ, η συγκίτρια είναι κατά, υπέρ. Η ομάδα του κυρίου Μπουσούτιλ, κατά, η λυπή, οι λυπές ομάδες, αποχές, το ΕΛΚ ψηφί. Απορρίπτεται. Η 10-20 της ΓΚΟΕ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 167 της ΑΦΕΤ, η συγκήτρια είναι υπέρ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1007 της ΓΚΟΕ, η συγκήτρια είναι κατά, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 508 των Πρασίνων, η συγκήτρια είναι κατά, υπέρ. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ωραία λοιπόν. Γκέραν. Ήθελα να πω στην ε, πολιτική μου ομάδα είναι ότι αυτή είναι η μόνη ψηφοφορία που δεν στηρίζουμε, δεν ακολουθούμε την εισηγήτρια. Ε... Κατανοώ ότι αυτή είναι μια ψηφοφορία για το Θιβέτ. Άρα η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιο είναι άλλο είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Η φιλελεύθερη, η πράσινη, η γκουε. Κατά παρακαλώ, οι υπόλοιποι. Ωραία. Κυρία εισηγήτρια, λυπούμεθα. Αλλά είναι μια... η πλειοψηφία είναι κατά. 182 ε, της ΑΦΕΤ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι άλλες δύο καλύπτονται. Η του Βαντέλεν είναι συμβατή. Η εισηγήτρια είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 4768 του Σούριαν. Η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ. Το έλκε. Και η κυρία Ανδρέασεν. Κατά. Η λυπή. Πλειοψηφούν. Αποχές απορρίπτεται. Η 47-65, ε, Η συγκήτρια είναι κατά. Υπέρ. Η ίδια κατά η ίδια πλειοψηφία αποχές, επίσης απορρίπτεται η 4362 του Γκουαλτιέρη. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Α, τότε θα πρέπει να γίνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 4362 του Γκουαλτιέρη. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν 40 παρόντες, 39 ε, ε, ψήφισαν, κάποιος κοιμάται. 18 ψηφί υπέρ, 21 κατά, δεν εγκρίνεται. 183 της ΑΦΕΤ, με μια προφορική τροπολογία. Θα πρέπει να διαγραφούν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Η σύγκριση είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται με προφορική τροπολογία 4453 του Βαντάλεν, με προφορική τροπολογία της ηγήτριας να αντικαταστούν τα 10% αυτής της γραμμής του προπολογισμού από το τμήμα αυτών των κονδυλίων υπέρ του, της τροπολογίας Βαντάλεν. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 184 της ΑΦΕΤ δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα μέτρα στο, ε, στον τομέα εργαλείου, σταθε, στο εργαλείου σταθερότητας. Η συγκίτρια είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά ε, το, εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Ε, το δεύτερο τμήμα υποστήριξη για μέτρα έως ότου συνδρομή προς τα θύματα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 185 της ΑΦΕΤ. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα καλύπτονται οι επόμενες Γαρίγα, Γκρέσλε και Αλβάρο. Η 4330 της κυρίας Κράτσα. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4454 του Βαντάλεν που είναι συμβατή αλλά η συγγήτρια είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 186 της Αφέτη. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4455 είναι συμβατή, αλλά η είναι κατά, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γερνάω τη σελίδα. 147 αφέτη. Η συμβήτρια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γαρίγα, Γκρέσλε, Πρόεδρος Άλβαρο, ευτυχής. 188 αφέτ. Η συγκίτρια είναι υπέρ, ποια είναι υπέρ. Κατά αποχές. 518 των πρασίνων. Ε, πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα του 518. Άρχεται η ψηφοφορία. Toujours. Ah, ça y est. Celui qui dormait s'est réveillé. 40 votants. 40 ψηφίσαντες. 13 υπέρ, 25 κατά. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Ε, και πάλι η τροπολογία της ΑΦΕΤ. Ψηφίσουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Γιατί το δεύτερο τμήμα καλύπτεται από το πρώτο τμήμα της προηγούμενης τροπολογίας την οποία υπερψηφίσαμε. Για το πρώτο τμήμα της ΑΦΕΤ η συγκίτρινη πέρι πέρι Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47-70 που είναι συμβατή. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά πλειοψηφία απορρίπτεται. 176 αφέτ. Η συγκίτρια υπέρ, είναι υπέρ. Κατά. Και ο Σουριάν είναι κατά. Abstention. Adopté. Αποχές εγκρίνεται. 190 αφέτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47-71 συμβατή, η συγκίτρια είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Το ΕΛΚ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 520 των πρασίνων που είναι επίσης συμβατή, αλλά η συγκίτρια είναι κατά, ποια είναι υπέρ. πράσινη και γκουε, κατά, οι άλλοι. Αποχές απορρίπτεται. 518 των Πρασίνων σε δύο τμήματα. Η συγκήτρια είναι υπέρ του πρώτου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, είναι η ίδια πλειοψηφία όπως και πριν, αλλά ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν της 518 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Reste un endormi. Il s'est réveillé. Le vote est clos. 14 pour 20. Τέλος της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Για d'autres votes 518 des Verts, ça sera la même majorité. Άρα θα έχουμε την ίδια πλειοψηφία και στα υπόλοιπα 518 των πρασίνων. Θα δούμε. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 191 ε, αφέτ. Η συγγήτη είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα καλύπτεται. Για τη 4456 Βαντάλεν. Η συγκήτρια είναι κατά του πρώτου τμήματος, αλλά το ψηφίζουμε τώρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συγκήτρια είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος, ποιοι είναι υπέρ, με προφορική τροπολογία που λέει αντικατάσταση του 10% από τμήμα του κονδυλίου, είναι λιγότερο ακριβής. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται 5-20 που είναι συμβατό αλλά η συγκίτρια δεν τη θέλει η υπέρ ποιοι είναι κατά συγγνώμη ξαναρχίζω λίγο ο πρόεδρος ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 αφέτ με προφορική τροπολογία που λέει να διαγραφεί το τουλάχιστον 30 εκατομμύρια. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5-20 των πρασίνων που είναι συμβατό αλλά η συγκίτρινη κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην επόμενη σελίδα. Έχουμε και πάλι ένα 5-18 των πρασίνων, οπότε υποθέτω πως έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, όλοι, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Δεύτερο τμήμα λοιπόν απορρίπτεται. 193 αφέτ. Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα γιατί το δεύτερο καλύπτεται και ο εισηγητής είναι υπέρ η εισηγήτρια με συγχωρείτε, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 194 ε, φέτη, η εισηγήτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44-58 βαντάλ είναι συμβατό με το 94, αλλά η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.53 ίντα. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44.59 φαντάλεν είναι συμβατό. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Η συντηρητική. Ποιοι είναι κατά. Ε, απορρίπτεται. 10.35 γκουε. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5.13 πρασίνων. Η εισηγήτρια εδώ αγαπά τους πρασίνους. Ποιοι είναι υπέρ κατά. Υπέρ κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν κατάλαβα ποιοι, ποιοι έχουν την πλειοψηφία. 5.13 των πρασίνων ψηφίζουμε κύριε Γενική Γραμματέα. Les collègues Les collègues votent. Il y en a un qui dort. Tant pis pour lui, on arrête le vote. Τέλος ψηφοφορίας. 20-20. Απορρίπτεται. Έχουμε τώρα την 5 19 Προτείνω να ψηφίσουμε αν μπλοκ όλες τις 519 για την επόμενη γραμμή, γιατί είναι συμβατές. Αν μπλοκ, αλλά σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 519, 19 εισηγήτρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Δεύτερο τμήμα της 519 υπέρ, κατά, να επαληθεύσουμε, αλλά νομίζω πως απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα του 519 ψηφίζουμε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Τα δεύτερα τμήματα των 19 απορρίπτονται. 42-23 Άρτογκ. Η συγκίτρια είναι κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 της Επιτροπής Ανάπτυξης, η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47-73 Σούριαν καταπίπτει, αλλά όχι 54 των γυναικών. Είναι συμβατές. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά... Αποχές. Εγκρίνεται. Sur le 5, les 519 qui arrivent. Για τις 519 που καταφθάνουν. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως καλύπτονται από την προηγούμενη ψηφοφορία, κυρία Συγχύτρια. Το δέχονται οι πράσινοι. Ωραία. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο με την 519 και φτάνουμε τώρα στο 4777 του κυρίου Σουριάν. Ε, η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Καλύτερα να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, δεν είναι απόλυτα σαφές. 47-77 Σουριάν. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Bon. D'autres se sont endormis. On arrête le vote, tant pis. 17 pour 23 contre, l'amendement est rejeté. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά. Ψηφίζουμε το επόμενο λοιπόν του κ. Σουριάν, τη 47-63, που η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Non, non, non, non, ils sont contre. Qui est contre. Κατά. Αποχές, η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Je suppose que c'est la même majorité tout à l'heure, mais enfin, je, je le soumets. La... 5-18 το πρασίνο πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 519 ισχύει η προηγούμενη ψηφοφορία. Είναι το το πρώτο τμήμα εγκρίνεται και το δεύτερο απορρίπτεται. Εντάξει. Φτάνουμε στην 171. Αφέτε. Και άλλες που είναι ταυτόσιμες, η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 196 αφέτ. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175 αφέτ. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. και η 876 που ήταν ταυτόσιμη, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε τη 4609 που είναι συμβατή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και ξεμπερδέψαμε την ε, κατηγορία 4. Au tout début de la liste de vote. Αναρχόμαστε στην αρχή του καταλόγου ψηφοφορίας με μια άλλη κατηγορία που είναι ευαίσθητη, που είναι η 1α. Bien. Mes chers collègues, pour Monsieur, Monsieur Lavia a demandé la parole. Ο κύριος Λαβία ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάτι σε σχέση με μια ψηφοφορία που έγινε. Όταν ετέθησε ψηφοφορία εκείνο το πακέτο για τις ειδικέ εκδηλώσεις, ε, όταν το ψηφίσαμε είπατε ότι μιλούσαμε για το σύνολο του πακέτου. Όμως από τη Γραμματεία καταλάβαμε ότι ψηφίσαμε μόνο κάποιες πρωτοβουλίες και όχι το σύνολο του πακέτου.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 η συγκίτρια εξηγεί, και εγώ το υπεθυπίζω και για τους υπόλοιπους, ότι για τα special events υπήρχε, υπήρξαν δύο συμβιβαστικέ. Η μία αφορά τα νούμερα που τα ψηφίσαμε unblock και μία συμβιβαστική που κάλυπτε όλες τις παρατηρήσεις που και αυτές ψηφίσαμε unblock και που αντικαθιστά τις παρατηρήσεις ε, και των τροπολογιών. Άρα, τώρα εντάξει, καταλάβατε. Oui. Naturellement, le compromis n'a pas repris, additionné toutes les... Αφού είχαμε συμβιβαστική, σημαίνει ότι αντικαθιστά τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στις τροπολογίες σας. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την κατηγορία 1α. Ψηφίζουμε για την 1α λοιπόν. Έχετε ένα ειδικό πίνακα για να απλοποιήσουμε επί τη βάση των συμβιβαστικών. Είστε έτοιμοι όλοι, το έχετε αυτό το πίνακα. Να ξεκινήσουμε ψηφίζοντας στην, το μπλοκ 1 που αντιστοιχεί σε τροπολογίες που ξεπερνούν το σχέδιο προϋπολογισμού. Και στη συνέχεια θα πρέπει να εξετάσουμε α, τροπολογία προς τροπολογία εκείνες που δεν αφορούν παρά μόνο τις πληρωμές. Για την υπομάδα λοιπόν 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στις τροπολογίες. τις μεμονωμένες για τη σειρά για τις διάφορες γραμμές με συγχωρείτε 020201 για τη γραμμή 020201 αυτό αντιστοιχεί στη σελίδα 6 του μεγάλου καταλόγου ψηφοφορίας η άλλη αποσύρει. Δεν είναι απαραίτητη. Alors, oui, madame, madame euh, oui. Jensen. C'était un split vote. Euh. Η κυρία Γένσεν, ήταν μια χώρα, Ψηφοφορία κατά τμήματα είχαμε ζητήσει και το αποσύρουμε. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσως την 323. Όχι. Όχι. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται για τον υποομάδα 1 φτάνει. Bon, donc, je comprends que sur la ligne 02, 02, 01, il n'y a plus lieu. Για τη 02, 02, 01 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Λοιπόν, για την 02, 04, 01, 02, που είναι στη σελίδα 12 της, του Γενικού Καταλόγου, υπάρχει μια τροπολογία της ΓΚΟΕ, που θα πρέπει να είναι η 933. και που αφορά μόνο τις πληρωμές. Πληρωμές. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Είναι υπέρ. Όχι, είναι κατά. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Η τροπολογία δεν είναι της ΓΚΟΕ. Είναι του ΕΛΚΑ. Υπάρχει το αίτημα της ΓΚΟΕ για χωριστή ψηφοφορία. Οπότε βλέπετε την ΚΟΕ αριστερά, αλλά επειδή ζήτησε κατά τμήματα πληρο... ψηφοφορία. Αλλά η τροπολογία είναι του ΕΛΚ. Ναι. Είναι η 777. Κοίταξε, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι θα ψηφίσουμε τώρα. Dans l'ordre. Bon. Bon, alors, je soumets au vote Λοιπόν, ψηφίζουμε λοιπόν, είμαστε στη σελίδα 12 του μεγάλου καταλόγου ψηφοφορίας. 02, 04, 01, 02. Είναι η γραμμή. Καταρχήν έχουμε την τροπολογία της ΓΚΟΕ για τις πληρωμές. Η συγγήτρια δεν τη θέλει. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, πάμε τότε στην 4686 που είναι πάλι της Γκουε. Η συγκίτρια δεν τη θέλει. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε τη 4580 Βέρτμαν. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε στην 777 όπου θα πρέπει να υπάρχει κανονικά πλειοψηφία. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, για τις πληρωμές περνάει η 777. Η Άλντε έχει αποσύρει την τροπολογία της για τη 040304, τη γραμμή 040304, που ήταν ένα αίτημα για κατατμήματα ψηφοφορία και περνάμε στην 080901 όπου η Γκούέ ζητά και πάλι χωριστή ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την 959 της ΓΚΟΕ και 4656 συγγύτερα είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ, κατά πλειοψηφία απορρίπτεται. Μπορούμε να πάμε λοιπόν άμεσα στην 785. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Εντάξει. Λοιπόν, για τις πληρωμές περνά εδώ η τροπολογία η συμβιβαστική. Πάει λοιπόν το μπλοκ 1. Τα ίδια θα κάνουμε τώρα για την δεύτερη υποομάδα. Καταρχήν ψηφίζουμε λοιπόν για τις υποχρεώσεις. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αλλά για τις πληρωμές υπάρχουν αιτήματα για ατοματική ψηφοφορία για δύο γραμμές. Η Άλντε ε, επιμένει, ναι, μάλιστα. Τώρα επιμένει. Πάμε στη σελίδα 26. À la page 26, et on est obligé de commencer par l'amendement και πρέπει να ξεκινήσουμε από την 713 των σοσιαλιστών. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Φτάνουμε στην τροπολογία 389. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι καλύπτει αυτό την γραμμή 040501. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Άλλη μια χωριστή ψηφοφορία μόνο για τις πληρωμές στη σελίδα 38 όπου έχουμε την γραμμή 080202 0202. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να το βρω. Έχουμε λοιπόν την 956 της ΓΚΟΕ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φτάνουμε στην 678, η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και έτσι όσον αφορά την πληρωμή αυτής της γραμμής, πληρωμές αυτής της γραμμής, τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε τώρα στην υπομάδα 3. Το ίδιο σύστημα. Καταρχήν να, ψηφίσουμε τη συμβιβαστική για τα νούμερα για την υπομάδα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αποχές. Όλη η πομάδα αυτή απορρίπτεται. mais Όμως πρέπει να ψηφίσουμε χώρια την τροπολογία των πρασίνων στη γραμμή 082001 που είναι στη σελίδα 55. Για το ίτερ. Ναι, πονηρούλιδες. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας που είναι οι υπαριθμόν... Δεν είπε ο πρόεδρος ποια είναι. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε θεωρούμε ότι οι πληρωμές αυτές είναι αυτές που αντιστοιχούν στην υπομάδα αυτή. Έχουμε και τώρα και κάποια υπόλοιπα. Τα λεφτοβέχς. Voilà. Alors, on n'a pas besoin euh, d'aller à la page, on peut se contenter de, de ce qui est sur le. Δεν, αρκεί, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, αλλά αυτά που είναι εδώ στον πίνακα. 02, 02, 08, 04, τροπολογία της Επιτροπής Μεταφορών, 77-13. Ποιοι συγκέντρες είναι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν ξε... ξέρω σίγουρα. 77-13. Φτάσαμε του 43. Ψηφίσατε όλοι. 21-21. Απορρίπτεται. Μία αποχή. Απορρίπτεται. 47-26 τώρα της Επιτροπής Προπολογισμών. Η είναι υπέρ. Υπάρχει το προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Με την προφορική. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία των γυναικών. 62-20. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ε, ποιοι είναι υπέρ. Η πράσινη και η γκουε. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία Ήτρε 6073. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8720. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τα σχόλια τώρα. Η τροπολογία 102 της Οικονομικής Επιτροπής. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Το έλεγε τι κάνει εκεί. Κατά είστε. Υπέρ. Ξανά υπέρ. Κατά. Τα αποχές εγκρίνεται. 814 υπέρ και η συγγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οπότε η 323 καταπίπτει και η επόμενη 43-39 395 Επιτροπή Επασχόληση υπέρ και η συγγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει 47-72 συμβατή η συγγήτρια κατά ψήφι υπέρ Τη 72 Το ΕΛΚ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Le... Le 400... Η 428. Καταπίπτει. 533 των πρασίνων εισηγήτρια υπέρ. Άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43-65 γκολτιέρι, συμβατή, εισηγήτρια υπέρ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 397 της απασχόλησης, εισηγήτρια υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 427 απασχόληση, εισηγήτρια υπέρ, υπέρ, κατά ηλεκτρονική υπολήθευση. Είμαστε στην 427. Άρχεται η ψηφοφορία. Ανοίξτε σας παρακαλώ την ψηφοφορία. Oh, oh. Όχι μυστική. Να ανοίξετε απλώς το μηχάνημα. Ξανά. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Πέρασε. Ισοψηφία 21-21 απορρίπτεται. 5-32 των πρασίνων. Εισηγήτρια υπέρ. Άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47-75 υπέρ. Εισηγήτρια υπέρ είναι. Κατά. Αποχές. Βιβλιοψηφία υπέρ εγκρίνεται. 43-63 Γκουαλτιέρη. Εισηγήτρια υπέρ. Άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 952 της ΓΟΕΣ, η τρεπέ. Contre. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Sur le 952 de la GUE. Για την 952 της Το Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά και όχι μυστικά. Πέρασα. 15 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται. 724. Εισηγήτρια υπέρ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4503 Βαντάλεν, εισηγητρία υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 277 Ήτρε, εισηγητρία είναι υπέρ. Κοντ, Κατά, αποχές εγκρίνεται. 4761 συμβατή υπέρ, εισηγητρία είναι κατά. Κατά, αποχές με την ίδια πλειοψηφία περίπτεται. 278. Επιτροπή Βιομηχανίας. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτεται και επόμενη. 43-58 Η Συγγήτρια υπέρ. Υπέρ. Ιστορική έρευνα. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές 7.25 7-25. Σοσιαλιστές. Ψήφι υπέρ. Και η συγγήτρια μαζί. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43-59. Γκουαλτιέρη. Συγκήτρια υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 726. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 528. Των Πρασίνων. Κατά πίπτη. Κατέπεσε. 529. Των Πρασίνων. Εισηγήτρια κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 775 του έλκης ή υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το επόμενο. Τα δύο επόμενα λοιπόν καταπίπτουν και ερχόμαστε στη 531 των πρασίνων. Η συγγήτρια υπέρ. Άλλη υπέρ. Κατά. Χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση εδώ. Διότι αυτά τα πυρηνικά μας έχουν οδηγήσει σε σχάση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Αυτή κι αν είναι πυρηνική σχάση στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. 8 υπέρ, 34 κατά. Παρακαλώ. Και καμία αποχή. Οπότε απορρίπτεται, μάλλον. 964. Γκουε. Συγκίτρια επίση υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά. Με την ίδια πλειοψηφία αποθέτω. Απορρίπτεται. 6.27 φιλελεύθερη συγγήτρια υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται όπως και η επόμενη. 41.65 του κυρίου Χάρτον καταπίπτει διότι εγκρίθηκε η συμβαστική. 727 με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 624 Η εισηγήτρια υπέρ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επόμενη. 966 γκουε για τον Ισραηλινό στρατό εισηγήτρια είναι κατά ψήφι υπέρ η γκουε και η πράσινη κατά. Κου, et les Πολλοί είναι κατά και οι σοσιαλιστές από αλλά η πλειοψηφία είναι κατά. Οι σοσιαλιστές δεν θέλουν να κατευθούν με αυτά τα στρατιωτικά ζητήματα. Επόμενη τοπολογία των Βρασίνων. Η υπέρ, άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 530. 114 έκον. Η συγήτρια υπέρ, άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και καλύπτει και την επόμενη. 112 για τους νέους πόρους. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και καλύπτει και την επόμενη. 113. Η ίδια ιδέα περίπου. Υπέρ, κατά. Αποχές, η ίδια 813 του ΕΛΚ. Εισηγήτρια υπέρ, άλλη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και καλύπτει και την εξωτερικών. 601 των φιλελευθέρων. Εισηγήτρια πέ Άλλη πέ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 973. Γκουε. Συμβατή με την προηγούμενη. Εισηγήτρια υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οπότε και ερχόμαστε στη Μαρή Κιουρί. 43-60 ψηφί υπέρ, εισηγητρία υπέρ. Κατά. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται η τοπολογία Γκολτιέρη. Συγγνώμη κύριε Πόρτος, τι θέλετε. Νομίζω ότι επιδείξαμε μια τροπολογία. Τη δική μου συγκεκριμένα. Όχι, είχε καλυφθεί, γι' αυτό δεν την ψηφίζουμε. Λοιπόν, 3.15 ε, της βιομηχανία. Δεν είναι καθόλου η Νταντίκ οι δύο προηγούμενες, η Γκούε και εγώ, αλλά όχι τα προηγούμενα, όχι τη Άλντε. Ναι, αλλά περίφθη, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ειλικρινά, πιστέψτε. 3.15 της βιομηχανίας, η ψήφη είπε και η συγκήτρια είπε κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για τους Ρωμά, 4.57 της Λίμπη, η συγκήτρια είπε είπε Σοσιαλιστές τι λένε. 4,57. Τίποτα δεν λένε οι σοσιαλιστές. Κατά. Αποχές. Δεν συμμετείχαν οι σοσιαλιστές, υπερψηφίστηκε. 5.35 ε, των πρασίνων. Gender budgeting. Συγκίτρια είναι υπέρ. Κατά. Για τον προπολογισμό των φύλων. Εντάξει, τα προπολογίσαμε και τα φύλλα και τα γέννη. Ψηφίσαμε την 1α, τελείωσε αυτό. Mes chers συνάδελφοι, κάντε λίγο ησυχία, γιατί θα πληρώσει η αντιπρόεδρος Χάουκ, θα φάει καμιά σφυριά εδώ πέρα. Είτε ο κύριος Δεάν ο οποίο αστείευεται για την κυρία Χάουκ. Ο κύριος Ντεάν θα την πληρώσει, όχι η κυρία Χάουκ. Λοιπόν. C'est très simple et très rapide. Πάμε τώρα στα πιλωτικά. Είναι πολύ απλό και πολύ γρήγορο και μετά θα έχουμε 5 λεπτά διάλειμμα για να συνεννοηθούμε για την ψηφοφορία για τα υπόλοιπα τμήματα, ιδιαίτερα για το Κοινοβούλιο. Εντάξει. Καλώς, πάμε. Στα πιλωτικά είμαστε τώρα. Έχετε ένα ξεχωριστό πάλι έγγραφο για τα πιλωτικά. Συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων πώς θα οργανωθεί η ψηφοφορία και σας προτείνω να κάνουμε blog μαζί μου όλες και για τα ποσά και για τα σχόλια. Γιατί στα πιλωτικά προγράμματα ε, παίρνουν ύπαρξη και σάρκα και οστά τα προγράμματα από τα σχόλια. Αλλιώ δεν υπάρχουν καν. Εκτό αν αντιταχθεί κανεί. Αλλά δεν μου φαίνεται λογικό να διαφωνήσει κανεί. Λοιπόν, ψηφίζουμε μαζί αυτό το έγγραφο που λέει πιλωτικά προγράμματα και αφορά και τα ποσά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις βεβαίως, όσο και τα σχόλια που επεξηγούν ε, το νόημα αυτών των σχεδίων. Υπέρ. Κατά. Abstention. Αποχές εγκρίνεται το σύνολο των πιλωτικών προγραμμάτων. Λοιπόν, τελειώσαμε το τμήμα 3, τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούμε να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Μπράβο σου, Φραντσέσκα. Bien. Alors maintenant, euh, Λοιπόν, σας προτείνω πέντε λεπτά διάλειμμα για να συνεννοηθούμε το πώς θα ψηφίσουμε τώρα τα υπόλοιπα τμήματα, τα θεσμικά όργανα. Λοιπόν, διακοπή λίγων λεπτών.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 ρωτήσαμε ήδη από την, ε, από την εισηγήτρια να μας πει ε, πώς επιθυμεί να, τους να μας πούν πώς επιθυμούν να ψηφίσουμε. Το γραπτό κείμενο σας έχει διανεμηθεί και θα προσπαθήσουμε συνεπώς να πάμε αρκετά αργά. Κανονικά θα μπορούσαμε να τελειώσουμε σε μία ώρα. Αλλά είπα στους συντονιστές ότι θα ήθελα, αν τελειώσουμε πριν από τις 12.30, να τους κρατήσω στην αίθουσα αυτή μαζί με τους διερμηνείς μέχρι τις 12.30, ούτε στο Ράιμερ Μπέγκε, ο οποίος ε, χθες το πρωί ε, στην αρχή της συνεδρίασής μας συνάντησε μια αντιπροσωπεία της πολωνικής ε, αντιπροσωπείας να μας ενημερώσει για το τι υπόθηκε ε, με την πολεμική Προεδρία. Ε, ε, Προβλήματα ΙΤΕΡ όσον αφορά την, τον προϋπολογισμό του 2012, για το οποίο εγκρίθηκε η γραμμή του προϋπολογισμού χθες. Λοιπόν, Όσον αφορά τους συντονιστές λοιπόν, να μην φύγουν μετά την ψηφοφορία γιατί θα πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση και να τοποθετηθούμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο τον πίνακα ψηφοφορίας και υπάρχει το κείμενο των προφορικών τροπολογιών που έχουν διανεμηθεί χθε το βράδυ σήμερα. Θα πάρουμε ε, το πίνακα 205 other sections, άλλα τμήματα. Θα ξεκινήσουμε για τις αποδοχές ε, για το, από το Κοινοβούλιο. Η 20.00 του, της, της εισηγήτριας. Η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ευχαριστώ. Αποχές εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίε τη γραμμή αυτή έχουν αποσυρθεί. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο κάπω ευαίσθητο που είναι τα, οι δαπάνες ταξιδίου και θέλαμε να γίνει μια ομού ψηφοφορία από κοινού. Ε, ε κύριε Σιγητά, πώς ε, επιθυμείτε να ψηφίσουμε αυτή την ε, κατηγορία δαπανών ταξιδίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να δώσω μια μικρή εξήγηση. Δηλαδή, για να έχουμε το μέγιστο βαθμό διαφάνειας, βάλαμε σειρά προς σειρά, αντιπαραθέσαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, τους ε, συμβιβασμούς που έγιναν στη συνδιαλλαγή, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και επετέθη με ένα συμβιβασμό στο Προεδρείο, αλλά υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες που δεν είναι πλήρως σύμφωνες με αυτό το συμβιβασμό και για να μην χάσουμε χρόνο θεωρώ ότι θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε τον κατάλογο της ε, ψηφοφορίας γιατί αν πάρουμε τις βασικές τροπολογίες θα, ε, θα δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση οι γραμμέ δηλαδή που καταπίπτουν λόγω, αυτής της, ε, λόγω αυτών των συμβαστικών τροπολογιών. Λοιπόν, σα προτείνω να ακολουθήσουμε τον κατάλογο. Λοιπόν, τα συνήθεια έξοδα ταξιδίου. Ο, ο κύριος Μποκρός ε, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια προφορική τροπολογία η οποία είναι σημαντική όσον αφορά το 1005 και το 1004. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να τις ψηφίσουμε. Ε, αν δεν έχετε το κείμενο, αν το έχετε, να το ψηφίσουμε. Αλλιώς θα ε, σας, το γραπα... θα διαβάσω. το έχουμε όσον αφορά την απολαύθερση του, δεσμα... του δεσμευτικού, του αποθεματικού, συγγνώμη. 15% να τεθεί στο αποθεματικό και εξετάζεται η εφικτότητα των μέτρων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών ταξιδίου, ούτω ώστε να γίνουν κάποιες προτάσεις για μελλοντικέ εξοικονομίες στον προπολογισμό. Ε, ε, περιλαμβάνει ε, flex economy ε, ταξίδια και την ε, αναθεώρηση των ρυθμίσεων σε σχέση με τις, ε, ε, την Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Προκρός. There Ναι, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια σημαντική προσθήκη όσον αφορά τη δικαιολόγηση. Την τελευταία φράση που λέει ότι δεν θα πρέπει, να γίνει αναπροσαρμογή όσον αφορά τις ε, δαπάνες ταξιδίου συμπεριλαμβανόμενων και των καθημερινών επιδομάτων. Ε, θα ήθελα να ψηφιστεί αυτό στην προφορική τροπολογία την οποία διαβάστηκε προηγουμένω. Τώρα, όσον αφορά τη μέθοδο ψηφοφορία, γιατί αυτό δεν αναφέρεται πλήρω στον κατάλογο ψηφοφορία και νομίζω θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια, να είμαστε ξεκάθαροι. Η πιο σημαντική τροπολογία είναι η τρίτη εδώ, η 2057 από τον εισηγητή, του εισηγητή του κυρίου Φερνάντες. Δεν έχουμε προβλήματα με τα ποσά, δεχόμαστε τα ποσά, δεχόμαστε τους αριθμούς, επίσης όσον αφορά αυτά που μπαίνουν στο αποθεματικό, αλλά θέλουμε να ψηφιστεί εδώ η προφορική τροπολογία αντί για τις παρατηρήσεις του εισηγητού και την, ε, και την αιτιολόγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν υπάρχουν πολλοί που ζήτησαν το λόγο. Λοιπόν, εκ μέρους του κυρίου Ποκρός και της ομάδος του θα υπάρξει μια προφορική τροπολογία για τη γραμμή αυτή του προπολογισμού που θα πρέπει να εξετάσουμε σε ε, όσον αφορά την τροπολογία 817. Ε, και την 10.05. Όσον αφορά τους σοσιαλιστές θα υπάρξει προφορική τροπολογία, υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τα ποσά, αλλά υπάρχει προφορική τροπολογία όσον αφορά τη θέση αποθεματικό και την τροπολογία 20.57. Ε, λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Αλβάρο, τη Χέλγα και μετά ε, τον Πόρτας. Ο κύριος Αλβάρο, ευχαριστώ πολύ σχετικά με την 2055 στην οποία αναφέρθηκε ο Γκέρεν, γιατί, 2057, ε, γιατί δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο. Εάν εγκριθεί η προφορική τροπολογία στην περίπτωση αυτή, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Δηλαδή, το τελευταίο τμήμα αναθεωρεί τους κανόνες όσον αφορά το ωράριο, θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά κύριε Πόκρος, όχι επειδή θέλω να το καταψηφίσω, αλλά επειδή ξέρω ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί ε, σε σχέση με το καταστατικό. Και θα ήθελα απλώς ε, να γνωρίζω κατά πόσο μπορούμε να πάρουμε τη σχετική απόφαση που περιλαμβάνεται στην ε, θεσμική συμφωνία στο καταστατικό, στον κανονισμό περιστατικής κατάστασης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτές τις παρατηρήσεις για το στο καθεστώς των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλβάρο. Ε, κατανοήσαμε ότι θέλετε, ότι θέλετε να γίνει χωριστή ε, ψηφοφορία. Η Χέλγα, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε, όπως είπε ο κ. Πακρός, αυτή την ε, χωριστή τροπολογία και θέλω να πω ότι στηρίζω τα όσα είπε ο Γκέρεν. Νομίζω ότι το κάνει πιο ξεκάθαρο όσον αφορά το περιεχόμενο και σε σχέση με τη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Έλγα. Αυτό μας κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Ο κύριος ε, Πόρτας έχει το λόγο. Η μόνη αμφιβολία που έχω εγώ είναι ότι το πρώτο τμήμα της παρατήρησης που έκανε ο συνάδελφος Γκόραν νομίζω πως είναι αντιφατική με την πρόταση της εισηγήτριας. Η συγγήτρια προτείνει το πάγωμα των δαπανών ταξιδίου συν μία μείωση 5% πέρα από την δημιουργία του αποθεματικού. Και η παρατήρηση του συναδέλφου Κόραν μιλά για πάγωμα. Πάγωμα δεν είναι μείωση, και γι' αυτό και νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να ψηφιστούν χώρια. Ε, συμφωνώ με τα όσα είπε δηλαδή ο συνάδελφο Άλβαρο, με τουλάχιστον ένα τμήμα. Ε, εγώ είμαι, συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκόραν, εγώ είμαι κατά όμως του παγώματος. Θέλω την μείωση 5% και το αποθυματικό του 15%. Α, ναι, και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Και εγώ έχω μια προφορική τροπολογία, αλλά είναι μετά. Να την εξηγήσω τώρα, την προφορική τροπολογία. Μα την δώσατε γραπτός. Ναι, αλλά είναι για άλλο σημείο. Να έχει διανεμηθεί, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Ο εισηγητή θέλει να πατήσει στον κύριο ε, Πόρτα, αλλά ο κύριο Βόγκαν θέλει να συμπληρώσει κάποια πράγματα. Ωραία, λοιπόν, Βόγκαν. Ντέρακ. Είμαι σίγουρος ότι ο εισηγητής θέλει να απαντήσει στον κύριο Πόρτας, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια αντίφαση, γιατί μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να περικόψουμε τη γραμμή του προπολογισμού κατά 5%, μπορούμε να το συμφωνήσουμε, αλλά επίση λέμε στι παρατηρήσει ότι πιστεύουμε ότι τα επιδόματα θα πρέπει να παγώσουν. Εδώ δεν υπάρχει αντίφαση. Μπορεί να γίνει η περικοπή αλλά μπορούν να, μπορεί να γίνει και το πάγωμα από την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για να περιπλέξουμε κάπως περισσότερο αυτή την ψηφοφορία. Αυτό που προτείνουμε οι σοσιαλιστές είναι τα σχόλια που, έκαναν, που έκανε ο Γκιόρεν, που είναι η αιτιολόγηση, να είναι τμήμα των σχολείων θα πρέπει να γίνει χωριστή ψηφοφορία, γιατί κατά πάσα πιθανότητα ορισμένε πολιτικέ ομάδε θα ψηφίσουν περισσότερο ένα τμήμα και θα καταψηφίσουν κάποιο άλλο. Όσον αφορά την ημερήσια αποσμίωση και την αναπροσαρμογή τους. Ωραία. Ο εισηγητής θα μας πει ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει και η στάση για την ψηφοφορία. Έχω την εντύπωση, αν κατάλαβα καλά, αλλά είναι κάπως δύσκολο, έχω την εντύπωση ότι όλες οι προφορικές ε, τροπολογίες που εξετάζουμε εδώ, που ανέφεραν οι διάφοροι παρβενέντες, εκτός από του, το, του κυρίου Πόρτας, αφορούν ε, την ε, τροπολογία 25, 25. Ε, και εδώ, ε, ε, κύριε Σιγητά, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα πει ότι, ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε τις ερωτήσεις νομικής φύσεως αλλά είμαι υποχρεωμένος και έχω και κάποιες αμφιβολίες εάν ε, μπορούμε στην αιτιολόγηση να κάνουμε κάποιες αλλαγές ε, κανόνων και να ζητήσουμε από το Προεδρείο, ε, να ζητήσουμε από το Προεδρείο. Διερωτώ και επίσης, γιατί αυτή είναι η πρώτη μου εδώ, εάν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε την αιτιολόγηση, εάν τις ψηφίζουμε εν γέννη, αλλά εδώ έχουμε μια νέα διαδικασία και τις ψηφίζουμε και ε, βάσει αυτού θα, θα ε, έχετε γίνει μια αλλαγή. Και τώρα όσον αφορά τα σχόλια, θεωρώ ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν. Αυτό το οποίο πρότεινα να γίνει μια περικοπή του 5% στη γραμμή αυτή των ταξιδίων υπήρξε μια τροπολογία των σοσιαλιστών που ήταν να παγώσει. Εγώ πρότεινα 15% να μπουν στο απαθηματικό και όλοι συμφωνούν. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία όσον αφορά την αιτιολόγηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το θέμα πολύ απλά και πιο στεναρά στο ψήφισμα. Και αν κάνουμε μια περικοπή της τάξης του 7% όλοι θα συμφωνήσουν στο Προεδρείο, δηλαδή 15% να μπει στο αποθεματικό εσώ το Προεδρείο παρουσιάσει μια μελέτη για όλες τις μορφές ταξιδίων. Θεωρώ ότι η δική μου τροπολογία καλύπτει την τροπολογία των σοσιαλιστών γιατί είναι ευρύτερη αυτή, γιατί και περιλαμβάνει όλους τους τύπους ε, ταξιδίων και οικονομίας. Και για τα άλλα θέματα υπάρχει το ψήφισμα και θα μπορούσαν ενδεχομένω να αληθούν μέσω του ψηφίσματος. Ε, ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι υποβάλλουμε μια προφορική τροπολογία και στη δική μου προφορική τροπολογία θα πρέπει να ψηφιστεί πριν από την τροπολογία του εισηγητού. Εάν αυτό ισχύει κάποια στιγμή, τότε, ε, κάποια μέρα, τότε δεν θα υπάρξει καμία απολύτω ε, τροπολογία. Δεν θα κατήθεται μια τροπολογία, θα ψηφίστηκε στη συνέχεια θα κατήθεται μια άλλη τροπολογία για να καταστρέφεται, να καταπίπτει η προηγούμενη τροπολογία και αυτό δημιουργεί τεράστια σύγχυση εγώ προσπάθησα ευθύ εξ αρχής να υπάρξει μια συνένεση. Ε, έστω και μετά την συμφωνία με το Προεδρείο στη Συνδιαλλαγή. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω σε τι χρησιμεύουν αυτές οι συνεδριάσεις της συνδιαλλαγής. Εγώ παρόλα αυτά πραγματικά έκανα μια προσπάθεια για να υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία. Και πιστεύω και το επαναλαμβάνω ότι στο ψήφισμα ε, θα είχαμε μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι στην αιτιολόγηση που τώρα θέλουν ε, να γίνει σχόλιο. Ε, καταλαβαίνω κύριε Σιγητά, αλλά θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση. Πράγματι προτείνατε εσείς ο ίδιος μία τροπολογία, εάν κατάλαβα καλά, που θα ήταν μία τροπολογία για την αιτιολόγηση ε, που θα γινόταν που θα αφορούσε Αυτά. τα συνήθεια έξοδα ταξιδίου. Λοιπόν, είτε θα κάνουμε ένα σχόλιο, είτε αυτό το οποίο μου φαίνεται πιο λογικό, θα προτείνεται να περιληφθεί στο ψήφισμα. Ε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια συνέντευξη μέσω του ψηφίσματος. Αυτό είναι που προτείνω εγώ και είναι αυτό το οποίο είχα ήδη προτείνει σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ωραία. Δηλαδή θέλετε να ψηφιστεί το κείμενο αυτό τώρα. Ε, νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει να περάσει το ψήφισμα ή όχι. Φυσικά. Ο Γκέραν έχει το λόγο. Συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνώ, γιατί νομίζω ότι χρειάζονται κάποια σχόλια για αυτή τη γραμμή του προπολογισμού. Τα χρειαζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε να ψηφίσουμε τα σχόλια. Αλλά συμφωνώ ότι κάναμε ένα σφάλμα, γιατί δεν προσθέσαμε τελευταία φράση τη αιτιολόγηση στα σχόλια. Και πραγματικά θα ήθελα να γίνει αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ένα απλό τρόπο να γίνει. Είναι οι πρώτες ε, δύο τροπολογίες που θα υπερψηφίσουμε τη θέση του εισηγητού για την περικοπή του 5% η 2057 θα υπερψηφίσουμε επίσης ε, τα ποσά αυτά. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το ψηφίσμα. Αν ε, ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτή είναι η συνήθι διαδικασία, να ψηφιστεί πρώτα το κείμενο, συμφωνούμε. Θα το καταψηφίσουμε και εάν καταπέσει θα ψηφίσουμε τότε την ε, προφορική τροπολογία. Ωραία λοιπόν, η Γιούτα έχω μία μικρή παρατήρηση για αυτό το οποίο έχει συνοψίσει ο Γκόραν. Δηλαδή την, να ψηφίσουμε την περικοπή του 5% και ταυτόχρονα όσον αφορά τα ποσά της τροπολογίας να, το, να αφήσουμε τα ποσά της 2057. Αλλά εδώ υπάρχει μια αντίφαση, γιατί έχουμε τα παλαιά ποσά και το αποθεματικό το οποίο έχει υπολογιστεί βάσει των παλαιών ποσών. Θα πρέπει να πάρουμε τα νέα ποσά που είναι περίπου 10 εκατομμύρια, δηλαδή είναι τα 5% των νέων, αριθμών, των νέων ποσών είναι περίπου 10 εκατομμύρια που θα πρέπει να μπουν στο αποθεματικό. Αλλιώ έχουμε ψηφίσει δύο πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Αλλά αφορά μόνο τα ποσά ή αν έχει το λόγο. Εγώ θα έλεγα όσον αφορά τις αρχές και χωρίς να μπούμε στην ουσία, πιστεύω ότι ο εισηγητής έχει δίκιο όταν λέει ότι δεν είναι δυνατόν ο καθένα να, διατυπώνει, να υποβάλει μια προφορική τροπολογία και να ζητείτε να ψηφίζετε. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε την τροπολογία, είπαμε ότι οι προφορικέ τροπολογίε θα πρέπει να ψηφιστούν εφόσον συμφωνεί ο εισηγητή. Αυτό είχαμε πει ω όρο. Μάλιστα κύριε Σιγητά. Κατανοώ αυτό το οποίο είπε ο Πόρτας και αυτό το οποίο είπε η Αντιπρόεδρός μας. Πιστεύω ότι η τροπολογία των σοσιαλιστών θα παγώσει και είναι αντίθετη η την τροπολογία που λέει ότι θέλουμε μια περικοπή της τάξης του 5%. Αγαπητοί συνάδελφοι, σταματάει εδώ η συζήτηση. Σας προτείνω να ψηφίσουμε γραμμή προς γραμμή οι δύο πρώτες γραμμές που αφορούν ε, το ποσό του αποθεματικού και αντίθετα υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για το σχόλιο. Δηλαδή καταρχήν το σχόλιο του εισηγητού θα ψηφίσουμε. Και αν και αν το σχόλιο του εισηγητού έχει την πλειοψηφία θα ψηφίσουμε τις άλλες προφορικές ε, τροπολογίες. Δεν υπάρχει αλλαγή στο σχόλιο. Ναι. Α, το ψηφίσουμε το σχόλιο. Ψηφίσουμε μάλλον επί του σχόλιο. Είναι οι τροπολογίε σου. Α, ξεκινάω από το δικό σου σχόλιο κάθε φορά. Λοιπόν, για την 2001 του εισηγητή. Δεν είναι η γραμμή, είναι η τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2069, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2057, αριθμοί. Και οι αριθμοί του αποθηματικού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σχόλια τώρα του εισηγητή. Δηλαδή, η όροι για την άρση του αποθηματικού. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορώ να ψηφίσω. Πριν από λίγο δεν μπορούσα. Όχι, δεν μπορώ. Πώς ακυρώνω. 45 <laughs> παρόντες και δύο που δεν ψηφίζουν. Ναι, εγώ είμαι. 17 <laughs> contre. 25 υπέρ, 17 κατά. Λοιπόν, υπερψηφίζονται τα σχόλια του εισηγητή και τα υπόλοιπα καταπίπτουν και τέρμα υπόθεση. Ναι, αυτό το πρόβλημα πάει, το ρυθμίσαμε. Άρα, μην ανησυχείτε, θα έχουμε κι άλλα για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε την ώρα μας. Έχουμε το ψήφισμα και να βρούμε συμφωνία... Και... Λοιπόν, 8-19. Α, όλα αυτά καταπίπτουν. Όλη σελίδα. Όλη σελίδα. γιατι 48-89 υπάρχουν παρατηρήσεις. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υποτίθεται ότι είναι συμβατέ. Όχι, είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται οι παρατηρήσει. Λοιπά έξοδα ταξιδίου. Το ίδιο πρόβλημα. Η προηγούμενη ψηφοφορία το ρυθμίζει το πρόβλημα. Έτσι νομίζω είναι το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα. Η ίδια ψηφοφορία. μάστε Ωραία, καλύπτεται. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στις ε, αποζημιώσει γενικών εξόδων. Τώρα θα ξεσπαθώσει ο Μιγγέλ Πόρτας. Ακριβώς. Εγώ είχα κάνει μία τροπολογία που πρότεινε μία συμφωνία για μείωση 25% στον τίτλο των γενικών ε, εξόδων των βουλευτών και τώρα η προφορική τροπολογία που κάνω ε, είναι αυτή η περικοπή να είναι απλά συμβολική. Δηλαδή να περιοριστεί στο 5% που δίνει μια εξοικονόμηση γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ και που είναι σαφές το ότι διακυβεύεται εδώ. Ε, οι βουλευτές δέχονται ή δεν δέχονται να αγγίξουμε άμεσα τα εισοδήματά τους. Είναι πρόταση του 5% και προτείνω να ψηφιστεί πριν από την πρόταση του εισηγητή, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα είναι μια τροπολογία για τους αριθμούς, για τα νούμερα. 5% της λοιπόν μείωση. Περιορίζουμε τη συζήτηση σε συμβολικό ζήτημα. Ακόμα μια φορά δεν πρόκειται εγώ να μπω μέσα στα θέματα νομιμότητας. Ο συνάδελφος Πόρτας είχε κάνει μια τροπολογία για το πάγωμα των μισθών ε, μετά αφού συμπεράναμε ότι ήταν παράνομο κάτι τέτοιο την απέσυρε, τώρα μιλά για 25% μείωση των γενικών εξόδων. Αντίθετα με αυτό που λέει ο, ο συνάδελφος Πόρτας, τα γενικά έξοδα δεν είναι μόνο, δεν είναι έσοδα των βουλευτών, είναι γενικά έξοδα για το γραφείο του Ευρωβουλευτή. Το πάγωμα ήδη είναι περικοπή και Εμεί ζητήσαμε το πάγωμα για να επιφύγουμε νομικά θέματα και το θέσαμε στο Προεδρείο. Εγώ, για παράδειγμα, έχω πολύ σοβαρέ εμβολίε ότι μια περικοπή 5% είναι κάτι το νόμιμο και δεν παραβιάζει το καθεστώ. Αλλά ακόμη μια φορά δεν θέλω να μπω εδώ στα νομικά ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά τη σειρά της ψηφοφορίας, δεν έχω πρόβλημα να γίνει εξαίρεση και να ψηφίσουμε πρώτα την πρόταση του συναδέλφου Πόρτας για αυτή εδώ την ψηφοφορία, Α, με την προϋπόθεση ότι όλα αυτά είναι νόμιμα, δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσουμε το... την πρόταση του κύριου Πόρτας πρώτα. Κανονικά ψηφίζεται πρώτα η πρόταση του Συγητή. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την κομψότητά του, διότι όντως ο κανόνας που ανέκαθεν εφαρμόζουμε στην Επιτροπή ε, των προπολογισμών και που εφαρμόζουμε και από χτε είναι ότι όταν υπάρχει τροπολογία του εισηγητή, ψηφίζουμε πρώτα την τροπολογία του εισηγητή και μετά ερχόμαστε στον, συνηθισμένο κανόνα με τη σειρά των τροπολογιών κτλ. Ε, δηλαδή τα πιο, τις πιο απομακρυσμένες τροπολογίες κτλ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε με τη συμφωνία του κύριου εισηγητή την ε, τροπολογία του κυρίου Πόρτας πρώτα. Κύριε Άρτον, ζητήσατε το λόγο. Όχι, ναι, ναι. Πέρα από τα διαδικαστικά ζητήματα, εγώ θέλω να στηρίξω οποιαδήποτε περικοπή γίνει σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, γιατί θα είναι ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα σε αυτούς τους καιρούς οικονομικής κρίσης. Μάστα. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα την τροπολογία 985 του κυρίου Πόρτας με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κύριε Ντουρά, απέχει. Μάστε. Ε, ερχόμαι λοιπόν στην τροπολογία του εισηγητή 20.03 και 20.75. Είμαστε στην 1006. Αποζημιώσεις γενικών εξόδων στην ε, σελίδα 252 του ελληνικού κειμένου. Λοιπόν, τροπολογία του εισηγητή υπερκατά Αχ, αποχές <coughs> εγκρίνονται. Οπότε, θεωρούμε πως όλες οι άλλες καταπίπτουν εκτός από τις παρατηρήσεις του κυρίου Βαντάλεν για την ε, πλήρη λογοδοσία. Α, έχουν αποσυρθεί. Α, με συγχωρείτε. Pouvons passer aux accidents. Oui, Monsieur Ellis. Euh, Μάλιστα, ο κύριος Έλλης, εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι για αυτές τις, ε, τα γενικά έξοδα δεν, είναι, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να τα δαπανίσουν όλα αυτά τα χρήματα, τα μέλη, μπορούν να τα ξαναβάλουν πίσω στον προϋπολογισμό. Ε, και αυτοί που τόσο πολυκόπτονται για το δημόσιο χρήμα, ας τα ξαναρίξουν πίσω στο κορβανά του Κοινοβουλίου. Χειροκροτήματα ακούω και από ό,τι καταλάβαμε ο James Ellis θα δώσει το καλό παράδειγμα πρώτος. Και εμείς θα τον ακολουθήσουμε. Εντάξει, James. 20.06 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Χονδρικά οι τροπολογίες του εισηγητή για τη Λισαβόνα συμφωνούν όλοι. Αν υπάρχουν τώρα άλλες θα σας το θυμισω 41.10 41-10 Ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 20-12 του εισηγητή. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέση αποθεματικό που ζητούν οι συντηρητικοί στην 875. Ο εισηγητής είναι κατά. Α, έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί. Περνάμε στο λοιπό προσωπικό. 2008 του εισηγητή ποιοι είναι υπέρ. Κατά. οι αποχές. πλειοψηφία είναι υπέρ, εγκρίνεται. Από εκεί και μετά οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Περνάμε στη γραμμή διερμηνής συνεδριάσεων. Και εδώ μπορούμε να ψηφίσουμε, ε, και εγώ μπορώ να ψηφίσω. 2067 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για τα νούμερα τώρα, οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Αντίθετα υπάρχει θέση στα στην 874. Ήδη έχει γίνει παρέτητη ενέργεια από το Προεδρείο, μπορούμε να την αποσύρουμε. Ισχύει και για την 827 και την 886. Καλύπτονται. Καλύπτονται. Ωραία. 2016 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου 2068 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Υπόλοιπη γραμμή, οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν. Α, συγγνώμη κύριο Πόρτας, αποχή. Α, είστε κατά, μάλιστα. La 41-12 euh, του κυρίου Άρτοξ στην επόμενη γραμμή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η Βαντάλεν έχει αποσυρθεί. 41-13 Αρτόγκ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Η Βαντάλεν έχει αποσυρθεί. 879 το συντηρητικών εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, σας ευχαριστώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επόμενη σελίδα. 41-14 άρτογκ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 900. Ε, ο συγκεκριτής είναι κατά, υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται είναι ταυτόσιμη με την επόμενη, οπότε ε, απορρίπτεται και αυτή. Φτάνουμε στην 826 που έχει αποσυρθεί και πάμε στην 885. Την έχετε αποσύρει πράσινη. Α, την έχετε αποσύρει και αυτή. Ωραία. «41-15 Χάρτογκ». Πέρκατα, αποχές απορρίπτεται. Η 836 έχει αποσυρθεί. 894 των πρασίνων διατηρείται. Διατηρείται το... Όχι, το αποσύρατε. Α, το αποσύρατε. 44-34 Βαντάλεν. Έχει αποσυρθεί επίσης. Διατήρηση συντήρηση κτηρίων. 831 έχει αποσυρθεί. 889 των πρασίνων έχει αποσυρθεί. Energy consumption. ενέργειας. Κατανάλωση ενέργεια. Το 2073 του εισηγητή υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Όλε οι υπόλοιπε καταπίπτουν για αυτή τη γραμμή. Ασφάλεια και επίβλεψη κτίριων. Δύο τροπολογίες αν μπλοκ του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Επόμενη γραμμή, 992 της ΓΚΟΕ, ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται, καθώς και οι επόμενοι. 10.43 υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά, κατά, αποχές, απορρίπτεται. <clears throat> Μεταφορικά μέσα. Ο κύριος Βαντάλεν δεν την έχει αποσύρει. Δύο τροπολογίες της Γκου. ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται και μπορούμε να περάσουμε στην γραμμή 2.30. Δύο τροπολογίες της Γκουέ ο συγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λοιπές δα... Απορρίπτονται. Λοιπές δαπάνες διοικητικές λειτουργίες. Δύο τροπολογίες της Γκουέ Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται γραμμή αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα. Τροπολογία του εισηγητή ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φαντάζομαι ότι οι υπόλοιπε καταπίπτουν όσον αφορά τα νούμερα, αλλά υπάρχει μια θέση αποθεματικό που ζητούν οι συντηρητικοί στην 878. Ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Στη γραμμή 302 υπάρχει η τροπολογία του κ. Φερνάντες, του εισηγητή, που δεν αφορά παρά μόνο τις παρατηρήσεις. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για τους αριθμούς 44-37 ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές νέα 9-20 ναι, ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επόμενο. Απορρίπτεται και αυτό γιατί το ταυτόσιμο. Τώρα για τις συνεδριάσεις 8-80 των συντηρητικών. Ο εισηγητής είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ο Βαντάλλαν την έχει αποσύρει. Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων. Γραφείου ταξιδίων. Τροπολογία άρτων 41-16 πέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8.33 έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία των πρασίνων 8.91 έχει αποσυρθεί. Ναι. Εντάξει μετά από πίεση του εισηγητή οι πράσινοι υποχωρούν. Αποσύρεται. 653. Άλντε. Τροφορική τροπολογία του εισηγητή. Είναι στον κατάλογο. Όχι δημιουργία νέας γραμμής, αλλά να τεθούν τα κονδύλια στην υφιστάμενη γραμμή. Έχουμε ήδη γραμμή για αυτά. Και προτείνω ότι δεν είναι κόμψο να έχουμε δύο γραμμές ε, για το ίδιο πράγμα, τον ίδιο σκοπό. Και προτείνω να βάλουμε στην παρατήρηση να βάλουμε αυτή την παρατήρηση που λέει αυτά τα κονδύλια και τα λοιπά για το κοινοβούλιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να μπει στη 3049 για αυτές την πίεση και για αυτές τις παρατηρήσεις. 3249 με συγχωρείτε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αυτό καλύπτει τις τροπολογίες DAF και εξωτερικών. Προχωρούμε. Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης. Το ελληνικό κείμενο είναι σελίδα 263. Έχει αποσυρθεί 2071. Και Σιγητά, να εξηγήσω, ε, γιατί το έχουμε συζητήσει. Αποσύρω την τροπολογία που ήταν για μελέτες του περίφημου πιλωτικού προγράμματος στα 2 εκατομμύρια και ζητώ να μπει ε, στο αποθεματικό εκτάκτον του contingency reserve αυτό το ποσό. Μάλιστα. Δεν αποσύρετε εσείς λοιπόν την τροπολογία σας. Ζητείτε ε, να ε, αλλάξει ε, γραμμή ενδεχομένως αυτό το κονδύλι και γραφή στον προπολογισμό για έκτακτα συμβάντα. Πάντως η Επιτροπή Εξωτερικών χάνει την τροπολογία της για να μην αλλάζουμε ε, τα νούμερα. Καταλάβατε όλοι τι ζητάει ο Μάλλον. Ε, έτσι όπως τροποποιήθηκε λοιπόν η τροπολογία την ψηφίζουμε. Ψήφι Και contre. Κατά. Νομίζω ότι χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Tiens, moi je suis toujours considéré comme... Εγώ θεωρούμε ακόμα υπεράριθμο. Α, voilà. Voilà, ça y est. Okay. Μάλιστα. Απεκατεστάθην. 44 είμαστε. Γιατί ψηφίζουν 40. Pardon, pardon. Ah, mais, mais, mais quel, quel vote Ας ψηφίσει. Χωρί Χωρίς ε, μικρόφωνο. Ξέρω, ξέρω, έχουμε έλλειψη σοσιαλιστών. Ναι, ναι, c'était moi qui en trop, il y Εγώ ήμουν υπεράριθμο, το έλκο, έχει σοσιαλιστέ. Essayez de voter. On va, on va, Προσπαθήστε να ψηφίσετε παρακαλώ να δω τι θα σα πει το μηχάνημα. Α, τώρα περσέβει ένας σοσιαλιστής. Bon, alors, euh, euh, abstenez-vous, abstenez-vous. Ψηφίστε αποχή για να το λύσουμε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, προχωρούμε. Πέρας ψηφοφορίες. 23 23 υπέρ 18 κατά. Άρα εγκρίνεται ε, η ε, τροπολογία του εισηγητού, καλά μία αποχή που είναι τη συναδέλφου μας σοσιαλιστών. Ερχόμαστε τώρα στο αποθεματικό της 8.38 για τις σχέσεις με το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εισηγητής δεν είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κατά του αποθεματικού. Άρα απορρίπτεται. Υπάρχουν όμως σχόλια. Ο εισηγητής είναι υπέρ των σχολείων. Ποιο είναι υπέρ των σχολείων σε αυτό το κονδύλι. Καταψηφίστε και το σχόλιο κύριε Σιγητά. Μάλιστα. Ψηφίζουμε όμως. Ο εισηγητή κατά. Ψήφι υπέρ. Του σχολείου. Κατά. Νομίζω ότι είναι πλειοψηφία υπέρ, αλλά ας το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να το ελέγξουμε. Η Χέλγα Τρίπελ. Ναι, χρειάζομαι λίγες εξηγήσεις για αυτά που ψηφίζουμε. Είμαστε στο 838 στα γερμανικά, τα και ο πρόεδρος. Πώς το λένε, 833, και εν πάση περιπτώσει 838 στα σχόλια, remarks. Και ο συγητής είναι κατά, σε διάφορες γλώσσες ο πρόεδρος. Αρχίζει ψηφοφορία. Και τώρα ουδής ψηφίζει. Πάλι μας περισσεύει ένα σοσιαλιστή. Αποχή. Πέρας. 17 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτονται και τα σχόλια. Μάλιστα. Προχωρούμε. Πιλωτικό έχει καλυφθεί. Συνεχίζουμε. 20-14 είναι το κονδύλι. Μισό λεπτό, πού είμαστε. page 228. Library expenditure. Non, non, mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Eh bien oui. Pas, oui, oui, c'est pas la ligne 2014, c'est amendement. Amendement, pardon, amendement 2014. Τροπολογία 2014, διορθώνει ο Πρόεδρος. Για τη βιβλιοθήκη. Και ψηφίζουμε για τα σχόλια. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου και όχι της Επιτροπής Προπολογισμών. Και για να διατηρηθεί η συμφωνία με το Προεδρείο και τα ποσά αποσύρω αυτή την τροπολογία και προτείνω 100.000 ευρώ να πάνε στο αποθεματικό για τα απρόβλεπτα και τα έκτακτα έξω. Μα είσαι σταλού, στο 2072. Ε, εγώ βλέπω ότι έχει αποσυρθεί. Ναι, το αποσύρω, αλλά κάνω προφορική τροπολογία. Ή στο κονδύλι, αν προτιμάτε. Η κυρία Ματέρα. Ναι, Πρόεδρε. Στο όνομα των υπογραφών των, της τροπολογίας 43-46 ε, αποσύρουμε αυτή την τροπολογία γνωρίζοντας πως ε, η υπόθεση αυτή είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου αλλά κυρίως γνωρίζοντας ότι το άνοιγμα αυτού στις θηρίδες θα έδινε ένα θετικό μήνυμα απέναντι στις προοπτικές και τις φιλοδοξίες ε, της Αραβικής Άνοιξης. Μιλώ εξ ονόματος όλων των υπογραφώντων την τροπολογία αυτή, 43-46. Με άλλα λόγια δηλαδή, κάποιοι συνάδελφοι Ιταλοί, τις οποίους υποστηρίζει και η κυρία Κρέσλε, ήθελαν να κάνουν μια τροπολογία για να χρηματοδοτήσουμε ένα γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Νάπολη για να λασάρουμε επαφές και πρωτοβουλίες ε, ε, σχέσεις με τις χώρες της ε, νότιας όχθης Μεσογείου. Ο εισηγητής ευαίσθητος αυτό το αίτημα και την τροπολογία έκανε άλλη δική του. Μετά από έντονες εντατικές διαβουλεύσεις μέχρι τα άγρια μεσάνυχτα με τους συντάκτες των τροπολογιών κατάλαβαν ότι δυστυχώς εμείς δεν είχαμε ούτε νομική βάση, ούτε καν πολιτική βάση, διότι δεν απευθυνθήκαμε στο Προεδρείο. Παράδειγμα, ο οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Αυτό είναι πολιτική απόφαση του Προεδρείου. Και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε με τη δημοσιονομική πτυχή που θα ψηφίσουμε. Αλλά ακόμα για αυτό το θέμα δεν υπάρχει απόφαση του Προεδρείου. Κατανοώ εγώ εκείνου που έκανα την τροπολογία και την κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα που ε, την αποσύρουν, την τροπολογία. Δημοσίως ανακοινώνει η κυρία Ματέρα την πολιτική πρωτοβουλία και υποθέτω ότι θα κάνει και ανακοινωθέν ε, δελτίο τύπου και θέλει το Προεδρείο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, Αν ασχοληθεί το Προεδρείο θα έχουμε πλέον και πολιτική βάση και νομική και ενδεχομένως ένα διορθωτικό προπολογισμό ή του χρόνου θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε. Εντάξει, κύριε εισηγητά, τούτων εκθέντων και λαμβανωμένων υπόψη, θεωρώ λογικό να αποσύρετε και τη δική σας τροπολογία. Έχετε το λόγο, δική σας είναι η τροπολογία. Μάλιστα, την αποσύρω όπως σας είπα και θα κάνω προφορική τροπολογία. Εδώ ή σε άλλο κονδύλι για τα απρόβλεπτα, το αποθυματικό, αυτές 100.000 και το συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε το Προεδρείο. Προτείνω όμως για να μην αλλάξουμε τα ποσά, όπως έκανα και στο θέμα ε, της Επιτροπής Εξωτερικών το περίφημο, αυτά τα 100.000 να μπουν στο αποθεματικό προβλέπτων και εκτάκτων. Contingency reserve λέγεται. Μάλιστα. Ζητήσατε το λόγο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 2072 του εισηγητού. Sous sa forme orale. Με αυτή την προφορική μορφή, εν πάση περιπτώσει. Δεν μιλάμε πια για την Άπολη, δεν γίνεται λόγος. Δυστυχώς την κρίμα. Ούτε το καπρί, καπρί σε φινί. Ε, Όπως έλεγε και το τραγουδάκι. Εν πάση περιπτώσει. Άλλες εποχές. Ψηφιπέ. Κατά. Α, τώρα θέλει μια ηλεκτρονική επαλήθευσούλα αυτό όμως. Μην ψηφίσετε εσείς παρακαλώ πάλι ε, σοσιαλιστές. Ε, έχουμε πάρα πολλούς σοσιαλιστές εδώ μέσα. Δεν τις χωράει τόπος. Εντάξει, πέρασε. 25 υπέρ, 16 κατά. Ούτως και αποφασίζεται με τον τρόπο που προτείνουμε. Συνεχίζουμε. Δημοσιεύσει με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα. 2059 του εισηγητού ψήφι υπέρ. Είμαστε σελίδα 265 στο ελληνικό κείμενο. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό τι σημαίνει ότι καταπίπτουν όλα τα υπόλοιπα για τα ποσά πάντα, για το ίδιο κονδύλι. Μάλιστα. Και θα περάσουμε στο επόμενο. 994 στην επόμενη σελίδα. Γκουε, εισηγητής κατά ψηφιπέ, αποχε αποχές, απορρίπτεται. 44-40 Βαντάλεν, εισηγητής κατά ψηφιπέ, κατά Κατά. απορρίπτεται. 8-82 συντηρητικό εισηγητής κατά ψηφιπέ, κατά Κατά. απορρίπτεται. 922 Ελευθερία και Δημοκρατία εισηγητής, κατά ψηφι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Καμία τροπολογία λοιπόν δεν εγκρίνεται στο κονδύλι αυτό. Επόμενο, Παρλαμεντάριουμ, 901, Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο εισηγητής κατά ψηφι κατά αποχές, απορρίπτεται. Επόμενη σελίδα, επόμενο κονδύλι. 9.95 της Γού, εισηγητής κατά ψηφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όπως επίσης και η επόμενη. Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων. 20-15 του εισηγητού. Αφορά μόνο τα σχόλια. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία της ΓΚΟΕ γιατί αφορά ποσά ο εισηγητή είναι κατά, 980 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 828, αν κατάλαβα καλά, έχει αποσυρθεί. Άρα θα ψηφίσουμε την 884 των συντηρητικών, ο εισηγητή είναι αντίθετο. ψήφι Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Επόμενη θέση του προπολογισμού. 80-83 των συντηρητικών ψήφι ο ή είναι κατά. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όπως επίσης λοιπόν και εκείνη του κυρίου Βαντάλεν. Επόμενη γραμμή του εισηγητού για τη Λισαβόνα 20.07. Ε, Είμαστε υπέρ υποθέτω τώρα συνθήκης Λισαβόνας, υπέρ κατά αποχές. Αυτά είναι απόρριες της συνθήκης και του Βαντάλεν καταπίπτει. Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. 41-17 Ο Εισηγητής κατά. ψηφι πέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44-44 Βαντάλεν. Ο εισηγητής είναι κατά. Ψήφι Έχει άλλα ποσά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 904 λέει ο πρόεδρος. 902 μάλλον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όπως και οι επόμενες που είναι ταυτόσιμες. Ερχόμαστε τώρα σε εισφορές ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Πάλι του κυρίου Χάρτον, 41-18, εισηγητής κατά ψηφί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44-45 Βαντάλεν έχει διαφορετικά ποσά, εισηγητής κατά ψηφί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 903 Ελευθερία και Δημοκρατία εισηγητής αντίθετος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όπως και τα υπολοιπα 2010. 20-10. Συνθήκη Λισαβόνα, εισηγητή, εγκρίνεται νομίζω, έτσι δεν είναι. Θεωρούμε ότι ψηφίσαμε ε, άπαξ και διαπαντό ό,τι έχει σχέση με τη συνθήκη Λισαβόνα. 982 γκουε. Ο εισηγητή αντίθετο, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Όπως επίσης και επόμενη. 20.04 Φυσίτου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στο περίφημο αποθεματικό για απρόβλεπτα. Εγκρίναμε κάποιες τροπολογίες σχετικές προηγουμένως για αυτά τα έκτακτα έξοδα και σας προτείνω αμπλοκ τώρα να ψηφίσουμε την 2008 ε, και 2004 υπέρ. Γιώραν, 2008 και 2004 είναι οι δύο τροπολογίες που ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Μιγκούε. Αποχές. Εγκρίνονται αυτές οι δύο τροπολογίες και τα υπόλοιπα πά κατά πίπτουν. Έμας. Η τροπολογία του εισηγητού. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην κατάσταση προβλέψεων, 2060 του εισηγητού ψήφι περ. Κατά. Το οργανόγραμμα μάλλον είναι αυτό. Ε, τέλειωσε το κοινοβούλιο. Δηλαδή τέλειωσε, εντάξει, το πληρώσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε την υπόλοιπη έκθεση Φερνάντες. 20-23 ε, του εισηγητού υπέρ για το δικαστήριο τώρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι υπόλοιπε. Ε, sur ε, le 20-24 του rapporteur, qui est pour. 24 Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Προσωρινές αποζημιώσεις. 20-26 του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για τις συντάξει 2027 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσωνή 2028 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2029 υπέρ του εισηγητού κατά αποχές εγκρίνεται δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων. 3.45 του εισηγητού. Μόνο τα ποσά. Υπέρ. Ορίστε. Όχι, δεν είναι του εισηγητού καθόλου, είναι των νομικών υποθέσεων. Γιούρι. Μου λένε ότι ο εισηγητή είναι υπέρ, αλλά βλέπω ότι είναι κατά. Τι θα γίνει. Υπέρ. Κανεί. Κατά. Όλοι. Εξαφανίστηκε. Προσωρινή πίστοση 20-30 του εισηγητή ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 3-31. Παροχές από εξωτερικού συνεργάτες στο γλωσσικό τομέα. Γιούρι, ο είναι κατά. Ναι, όχι, ναι, κατά είναι. Ψήφι πέ, κατά. Η πλειοψηφία χαίρεται. Επαγγελματική επιμόρφωση. Γιούρι, ο εισηγητή είναι κατά. Υπέρ της 332, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού. Ο εισηγητή είναι κατά τη τροπολογίας αυτή. Υπέρ. Contre. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, οι τροπολογίες 2031, 2032, 2033 του εισηγητού έχουν απαλληφθεί. Εν πάση έχουν αποσυρθεί εννοώ. Έτσι δεν είναι. Ερχόμαστε λοιπόν στην 2035, αγορά εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και λογισμικών. 2035, ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενο κονδύλι εξωτερικές ε, συνεργασίες κτλ. 2036 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο. 3.36. Εισηγητής κατά ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίφτεται. 3.37. Πάντα νομική επιτροπή και πάντα αντίθετος εισηγητής. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.38 υπέρ. Ο εισηγητής είναι κατά ψήφι υπέρ. Κατά. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 3.39 γιούρι το ίδιο. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 3.40 γιούρι τα ίδια. Η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 3.41 γιούρι το ίδιο. Η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. δημοσίευση γενικού χαρακτήρα. 2034 έχει αποσυρθεί. Η 342 των νομικών θεμάτων. Τα ίδια ισχύουν, ίδια αποτελέσματα, ίδιες πλειοψηφίες απορρίπτεται. Τα δικαιώματα τώρα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων. 2038 του ψήφι Π. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αποδοχές και αποζημίωση. 2061 του ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 2020 τοπολογία. Όπως λέμε Ευρώπη 2020 αυτό. Ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε και διεκπεραιώνεται αυτό το κονδύλι. Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα. 20-22 εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και καταπίπτουν οι υπόλοιπε για το ίδιο κονδύλι. Λοιπό προσωπικό 4104 Χάρτονγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με την πλειοψηφία. Διάφορα 4614 Βέρτμαν υπέρ. Κατά αποχές έχουμε πλειοψηφία κατά. Διερμηνή συνεδρία 2021 του κυρίου Φερνάνδης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και καλύπτεται το κονδύλι έτσι. Ερχόμαστε στην Επιτροπή Περιφερειών. Αποδοχές. Κύριε Σιγητά, έχετε αποσύρει την τροπολογία σας, μάλιστα. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία χάρτων 4101. Ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν προσωπικό, άλλη τροπολογία χάρτων, 4102, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Υπηρεσίες Διερμηνίας της Επιτροπής Περιφερειών, 2040, Φερνάντες, ψήφι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και διεκπαιρώνεται έτσι το κονδύλι. Επαγγελματική επιμόρφωση 2037 του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καθαρισμός και συντήρηση. 2041 του εισηγητού είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατανάλωση ενέργειας 2042 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ασφάλεια και επίβλεψη κτίριων 2043 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 2062 έχει αποσυρθεί, έτσι δεν είναι κύριε Σιγητά, μάλιστα. Ανάθεση υπηρεσιών 2044 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. θηλεπικοινωνίες 2045 του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 844 των σοσιαλιστών. Α, όχι, έχει καλυφθεί αυτό. Ε, αποδοχές και επιδόματα. 2063 υπέρ. Είμαστε στο διαμεσολαβήτη τώρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεδριάσεις γενικά. 2048 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επικοινωνία και δημοσιεύσεις. 2047 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε φτάσει στον Ευρωπαίο Υπόπτη Προστασίας Δεδομένων. 2050 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2064 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τροπολογία του κυρίου Χάρτον 4107 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Alors, sur le 197, 197. Τι προτείνει ο εισηγητής εδώ? Προτείνω γιατί ε, οι όροι για το αποθεματικό έχουν πληρωθεί. Ε, προτείνω λοιπόν να ε, δεχτούμε το ποσό και να άρουμε το αποθεματικό. Άρα εγγράφονται στη θέση του προπολογισμού αυτά τα ποσά. Δηλαδή στο σχέδιο είναι στο αποθεματικό και τώρα δίνεται να μπει στον κανονικό προπολογισμό, στη γραμμή. Υπέρ, κατά, αποχές. Οπότε έχει εγγραφεί το ποσό αυτό ε, στη γραμμή του προπολογισμού. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο κονδύλι 4107 χάρτον. Ο συγητής κατά ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επόμενο κονδύλι. 4107 πάλι χάρτονγκ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η Ελευθερία και η Δημοκρατία έχει δύο τροπολογίε. Εισηγητής κατά, ψήφι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 198 νομίζω ταυτίζεται με την τροπολογία του εισηγητού. Δηλαδή, στο σχέδιο του προπολογισμού υπάρχει ένα αποθεματικό, προτείνει να διατηρηθεί το ποσό αλλά να εγγραφεί στη γραμμή του προπολογισμού. Μάλιστα, ε, επαναφέρουμε το σχέδιο προπολογισμού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κοινωνική κάλυψη. Τροπολογία χάρτων 4107. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άλλο χάρτον 4107 για το επόμενο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασιούχοι. Το ίδιο είναι για το πόσο πάλι να φύγει από το αποθεματικό και να έρθει το ίδιο ποσό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει και με τη 200. Όχι, όχι. Είστε αντίθετος. Ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Γκολτιέρη. Για τη 200. Ναι, για τη 200. Είναι και αυτή μια τροπολογία της Επιτροπής Εξωτερικών. Εμείς είμαστε υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά αλλά ζητούμε ως προφορική τροπολογία να αρθεί το αποθεματικό. Και μετά θα ψηφίσουμε διαφορετικά μεταξύ μας. θα ψηφίσουμε και όπως και στις προηγούμενες τροπολογίες που βάλαμε το ποσό αυτό στην κανονική θέση του προπολογισμού και όχι στο αποθεματικό. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Vous êtes en faveur de... είστε υπέρ της απολογίας 200. Και ο εισηγητής είναι κατά. Ψηφίζουμε τη 200. Oui, oui. Χωρίς το αποθεματικό. Madame Jensen. Κυρία Jensen. I'd, I'd like to ask the question again. Who is making oral amendments here? Θέλω να ρωτήσω και πάλι ποιος κάνει οι προφορικές ε, τροπολογίες. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εισηγητή αν την αποδέχεται, γιατί θεωρώ ότι έχουμε έναν κανονισμό που λέει ότι ο εισηγητής είναι αυτός ο οποίος υποβάλλει προφορικέ τροπολογίε. προφορικές τροπολογίες. Έχετε δίκιο. Κύριε εισηγητά, χωριστή ψηφοφορία. Λοιπόν, με άλλα λόγια, προτείνεται να ψηφίσουμε καταρχήν το ποσό και στη συνέχεια το αποθεματικό. Ωραία λοιπόν. Δεν είναι προφορική τροπολογία. Ωραία λοιπόν. Άρα είμαστε σύμφωνοι. Μιλάμε για την 200. Μιλάμε για την τροπολογία περιθμών 200. Λοιπόν για τη 200. Για το ποσό. Ποια είναι η θέση του εισηγητού. Ε, το ποσό για να αποκατασταθεί το σχέδιο προπολογισμού και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε το αποθεματικό. Θα το ψηφίσουμε μετά. Αν δεν ε, ψηφιστεί το ποσό δεν υπάρχει κάτι που να πει στο παθηματικό. Ωραία λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ. Υπέρ του ποσού. τη 200. Κατά. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, του ΒΕΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπάρχουν τέσσερις που δεν έχουν ψηφίσει. Πέρα στις ψηφοφορίες, 18 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι κατά. Άρα απορρίπτεται αυτή η τροπολογία υπαρθών 200. Ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε το αποθεματικό. Όχι. Δεν υπάρχει πλέον, ε, δεν έχει νόημα το αποθεματικό. Λοιπόν, ίδια κατάσταση για τη 201. Ωραία. Ίδια ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ευχαριστώ. Άλλαξε κανείς. Όχι, είναι η ίδια πλειοψηφία. Άρα λοιπόν απορρίπτεται επίσης. Άρα θα περάσουμε στην ε, τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών 2066 του εισηγητού υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. 2066 του εισηγητού που φαίνεται ότι γύρει μεικτά συναισθήματα. Λοιπόν, ηλεκτρολογική επαλήθευση είναι η ώρα του απεριτήφ, αλλά ακόμα έχουμε κουράγιο. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορία. 17 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Η 4108 του Χάρτονγκ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Για τη 202 τώρα. είναι και πάλι μια νέα επιχείρηση του Γκουαλτιέρη. Όχι, κύριε Σταγητά, ισχύει το ίδιο όπως και πριν. Άρα η ίδια πλειοψηφία. Ο κύριος Φερνάντες τώρα είναι υπέρ. Ωραία λοιπόν. Άρα αποκαθίστατε το σχέδιο του προπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά για το ποσό. αποκατάσταση κατάσταση σχεδίου προπολογισμού υπάρχει μια πλειοψηφία. Τώρα, ε, προτείνεται να μπει στο αποθεματικό. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Καταργείται. Όχι, δεν το προτείνει κανείς. Λοιπόν, για την άρση του αποθεματικού εφόσον στην τροπολογία προβλέπετε το αποθεματικό θα το ψηφίσουμε. Ο εισηγητής ε, προσχώρησε στα επιχειρήματα σοσιαλιστών για την άρση του αποθεματικού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές, άρα όχι στο αποθεματικό. Αντίθετα, για, το 42, για την 4296 προτείνεται αποθεματικό από την κυρία Γκρέσλε. Ο συγκητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ του αποθεματικού, της θέσης αποθεματικού. Κατά. Alors, vote électronique pour savoir... Ηλεκτρονική επαλήθευση για να δούμε για το αποθεματικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. 2.500.000 ε, μπαίνουν στο αποθυματικό. Στη συνέχεια θα, μπούμε, ε, θα περάσουμε στην επόμενη, σαν 1.08 του Χάρτον. Υπέρ, κατά, α, αποχές απορρίπτεται. Η 203, η 203 τώρα, θα ψηφίσουμε καταρχήν τις πιστώσεις. να αποκατάσταση του σχεδίο προπολογισμού. Ποιος είναι υπέρ του ποσού. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τα ποσά. Της 203 ε, για τα έπιπλα. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. 20 προς 20 απορρίπτεται. Άρα θα ψηφίσουμε το αποθεματικό εφόσον δεν υπάρχει φύση πλέον τροπολογία. Τώρα, γραμμή 210-4108 του κυρίου Χάρτογκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 213-4108 του κυρίου Χάρτογκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη γραμμή μόνο 204 τη Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Βρισκόμαστε ενώπιον του ιδίου προβλήματος. Καταρχήν όσον αφορά την αποκατάσταση του σχεδίου προπολογισμού υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Βρισκόμαστε στη 204 για το ποσό του σχεδίου προπολογισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 20 κατά. Δεν υπάρχει αποκατάσταση προπολογισμού, άρα δεν μπαίνει τίποτα στο αποθεματικό. Τώρα για την 205 η ίδια, θέση, ίδια τοποθέτηση, η ίδια πλειοψηφία. Εάν κάποιος θέλει να αλλάξει γνώμη, παρακαλώ να το δηλώσει. Για την 206 τώρα, ίδια κατάσταση. 207 το ίδιο, η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 210 ιδία κατάσταση. Η ίδια τοποθέτηση, η ίδια πλειοψηφία προκειμένου να απορριφθεί. Άρα στη συνέχεια έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, έχει καλυφθεί. Θα περάσουμε στη γραμμή 3051 του εισηγητού. Υπέρ παρακαλώ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Γιατί εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων. 2051 ψηφίζεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. 16 23 κατά απορρίπτεται. Άρα είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω σε ψηφοφορία της αδέρμεδρανή του κ. Χάρτογκ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα φτάνουμε στην 209. Καταρχήν για τα ποσά. Στη συνέχεια για το αποθεματικό. Για το ποσό, για τα ποσά ποια είναι η γνώμη σας κύριε Σιγητά. Για την τροπολογία υπαριθμών 209. Ε, συγητής, ε, ναι, αποδέχομαι το ποσό και προτείνω τα 5 εκατομμύρια που αφορούν την γραμμή 3.000 και τη 3.003. Ε, αυτές αφορά η τροπολογία υπαριθμών 209 και λέω ότι 5 εκατομμύρια θα πρέπει να αποδεσμευθούν ως επίσημη, ε, καθώς ελέγχθη επίσημη απόφαση να υπάρξει μια αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, καταρχήν, για τα ποσά και στη συνέχεια θα δούμε τι γίνεται με το αποθεματικό. Για να αποκαταστήσω το σχέδιο προπολογισμού, η είναι υπέρ. Ποιο άλλο είναι υπέρ. Παρακαλώ, κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Άρα λοιπόν εγγράφεται αποκατάσταση του σχεδίου προπολογισμού. Τώρα, όσον αφορά θέσεις αποθεματικό, στην ε, τροπολογία προτείνεται εκεί, προτάθηκε. Εκεί όπου είχε προταθεί να μπουν στα αποθεματικά 13.300.000, αν κατάλαβα καλά, βάζουμε στο αποθεματικό 5 εκατομμύρια μόνον, διευκρινίζοντας ότι θα δοθούν στην αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Λοιπόν, ε, ποιος είναι υπέρ αυτής της πρότασης. Le, Ο εισηγητής προτείνει να μπουν στο αποθεματικό 5 εκατομμύρια και όχι 13,5 αλλά 5 μόνον εκατομμύρια που είναι τα 5 εκατομμύρια τα οποία προορίζονται Πέντε εκατομμύρια λοιπόν τα οποία προορίζονται στην αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ποιος είναι υπέρ αυτής της θέσης απαθηματικό. Όχι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Κύριε Σεϊτά, έχετε πάλι το λόγο. Έκανα μια τροπολογία για να προσπαθήσω όπως πάντα να πετύχω κάποιο συμβεβασμό. Και πίστεψα ότι οδεύω προς έναν συνολικό συμβιβασμό, αλλά αυτή, τη στιγμή έχουν έτσι τα πράγματα, αποσύρω την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, θα βάλουμε στην τροπολογία την τροπολογία που βάζει στο αποθεματικό 13,5 εκατομμύρια τότε, ε, συνεπώς λέει ο πρόεδρος. Έχουμε ήδη αποκαταστήσει το ποσό του σχεδίου προπολογισμού. Αλλά η τροπολογία περιλάμβανε την αποκατάσταση του σχεδίου προπολογισμού και τη θέση αποθεματικών των 13,5 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν ψηφίζουμε τα 13,5 εκατομμύρια αποθεματικό. Υπέρ. Κατά οι σοσιαλιστές που όμως είναι απομονωμένοι. Άρα, άρα δεν μπαίνουν στο αποθεματικό. Υπάρχει αποθεματικότητα τη εκατομμύρια. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Η τροπολογία εγκρίνεται. Άρα αυτά τα 13,5 εκατομμύρια μπαίνουν στο αποθεματικό. Ωραία, λοιπόν. Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω. Τέλο. Ε, Φτάνω προ το τέλο. 4109 του κυρίου Χάρτογκ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Βιάστηκα. Το εξωτερικό προσωπικό. 2053 ε, του εισηγητή του υπέρ 2053 υπέρ κατά θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση για την 2053. Άρχεται η ψηφοφορία. Votez, votez, votez. Le vote est λοιπόν πέρα τη ψηφοφορία. Αποτέλεσμα. 20 ψήφοι πέρα 19 κατά εγκρίνεται η τροπολογία. Άρα η επόμενη καταπίπτει τώρα η 209. Δεν χρειάζεται πλέον να ψηφίσουμε το ποσό, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουν το αποθεματικό. Έτσι δεν είναι κυρία Σιγητά. Ναι, είναι το ίδιο. Άρα καλύπτεται. 2053 καλύπτει όλη τη γραμμή. Άρα λοιπόν θα περάσουμε στην 3002. Η 2054 του κυρίου Φερναντές. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος άλλος είναι υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον είναι η ίδια πλειοψηφία με την προηγούμενη. 2054. Άρχεται ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρασε τη ψηφοφορίας. 21 points. 21 ψήφοι υπέρ, 19 κατά και πάλι μια μικρή πλειοψηφία. Άρα καταπίπτει. Καταπίπτουν και οι λοιπές. Η επόμενη γραμμή 3.03, 2052 του εισηγητού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές είναι η ίδια πλειοψηφία. Κανείς δεν άλλαξε γνώμη, άρα εγκρίνεται και άρα καταπίπτουν και οι υπόλοιπε. Τώρα για τη 30.04, 25 ε, του υπέρ. Κατά, η ίδια πλειοψηφία επίση, δεν άλλαξε κανεί εντωμεταξύ γνώμη, άρα εγκρίνεται. Οι λοιπέ καταπίπτουν. Τώρα ήρθαμε στη 41.09 του κυρίου Χάρτονγκ, υπέρ κατά, ευχαριστώ, απορρίπτεται. Τώρα ερχόμαστε τελευταία γραμμή 2065 του εισηγητού. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τελευταία τροπολογία για το οργανόγραμμα ίσως θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ, τελειώσαμε. Αλληλούια. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ λοιπόν και θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής και εγώ ε, θα κάνουμε μικρή ανακοίνωση τύπου στις 2 η ώρα για να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα και χαίρομαι για αυτό το αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά τιμά την Επιτροπή Προπολογισμών η οποία πέτυχε να εξεύρει την ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας σοβαρότητας που επιτάσσει η κατάσταση και της ε, φιλοδοξίας. Λοιπόν, αποδεσμεύω τα μέλη της Επιτροπής και τους ε, ακροατές που δεν ε, είναι μέρος της Επιτροπής των Συντονιστών που θα συνεδριάσουν σε λίγο θα ψηφίσουμε το ψήφισμα στην συνεδρίασή μας στις 11 Οκτωβρίου. Το ψήφισμα θα ψηφιστεί στις 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν, για δύο λεπτά διάλειμμα.